Καλησπέρα σας. Ξεκινάμε το σημείο 16, παρουσίαση των προτεραιοτήτων της Εστονικής Προεδρίας στον τομέα της δικαιοσύνης. Θα ε, καλωσορίσω τον Υπουργό Δικαιοσύνης ε, της ε, Εστονίας. Χθες είχαμε ε, τον Υπουργό Εσωτερικών με τον Υπουργό Εσωτερικών είχαμε συναντηθεί στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνη και Εσωτερικών Υποθέσεων ε, και καλύψαμε πολλά ενδιαφέροντα θέματα όπως η ηλεκτρονική ε, δικαιοσύνη, ε, η εν μέρη χτες καλύψαμε και το θέμα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας και άλλα ζητήματα που άπτονται της δικαιοσύνης. θα δώσω το λόγο λοιπόν τώρα στον Υπουργό Δικαιοσύνη για να μας ε, ε, κάνει την παρουσίασή του και μετά θα περάσουμε σε ερωτήσεις και απαντήσεις. Ο κύριος Ρέινσαλου. Καταρχήν θα μιλήσω στην, ε, στα ιστονικά. Είναι μεγάλη μου τιμή να βρίσκομαι εδώ σήμερα ε, για να σας παρουσιάσω τις προτεραιότητες της Προεδρίας μας σε αυτήν την πολύ σημαντική επιτροπή. Κύριε Πρόεδρε, η Εστονία θέλει να υιοθετήσει μία ε, πολύ ρεαλιστική προσέγγιση με υλοποιήσιμους στόχους ε, καθ' όλη τη διάρκεια της Προεδρίας της και θέλουμε να πετύχουμε μια σειρά στόχων σε μια σειρά ζητήματα. Εξετάζοντα τι προτεραιότητε στον τομέα τη δικαιοσύνης. Ξεκινώ ε, με την ε, πολιτική στο ποινικό δίκαιο. Υπάρχουν πολλά εκκρεμή ζητήματα. Ε, καταρχήν το θέμα του, της Ευρωπαϊκής Θα επανέλθω σε αυτό αργότερα, στο τέλος της ε, ε, παρουσίασής μου, για να σας παρουσιάσω την, πρώτη, την θέση του Συμβουλίου. Ε, πολύ συνδεδεμένο θέμα έχει, είναι το προσχέδιο κανονισμού για το, τη Eurojust, το οποίο ε, τελούσε σε ύπνωση για κάποιο καιρό, ε, αλλά τώρα ε, έχει ξαναξεκινήσει. Το Συμβούλιο έχει έχει ολοκληρώσει σχεδόν όλες τις συζητήσεις κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της Λετωνίας το Μάρτιο του 2015. Η Μαλτέζικη Προεδρία επίση ολοκλήρωσε συζητήσεις για την ε, Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το Συμβούλιο αυτή τη στιγμή τελειώνει κάποια ε, τελευταία θέματα ε, ευθυγραμμίζοντας το καθεστώς προστασίας των δεδομένων με το καθεστώς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις με το Κοινοβούλιο το, μόλις το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθετήσει την θέση του. ελπίζω να προχωρήσουν γρήγορα οι τερμερείς διάλογοι. Δεύτερον, ε, η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και άλλων σοβαρών ε, εγκλημάτων είναι επίση σημαντικό πρόβλημα. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι τα χρήματα που έρχονται από εγκληματικέ δραστηριότητε δεν θα πρέπει να χρηματοδοτούν άλλα εγκλήματα. Ε, η οδηγία για την αντιμετώπιση της νομοποίηση παράνομων προσόδων μέσω του ποινικού δικαίου και της αμοιβή αναγνώρισης θα είναι ψηλά στη μέση διάταξη. Ε, Επίση, υιοθέτησε το Συμβουλίο τη Γενική Προσέγγιση για την Οδηγία για την Καταπολέμηση ε, τη ε, νομοποίηση παρανόμων εσόδων μέσω του ποινικού δικαίου. Ελπίζουμε το Κοινοβούλιο θα συμφωνήσει το συντομότερο ότι είναι σημαντική προτεραιότητα και θα συνεργαστούμε ε, σε αυτό το ζήτημα κατά τη διάρκεια τη Προεδρία μα. Η Προεδρία επίση έχει ω στόχο να καταλήξει μια γενική προσέγγιση για την πρόταση περί κανονισμού για την εμβαία αναγνώριση ε, ε, της, ε, των ε, ενταλμάτων ε, δέσμευσης ε, και δήμευσης μέχρι το τέλος του χρόνου. Όπως ξέρετε η Κομισιόν υπέβαλε μια πρόταση κανονισμού για πρώτη φορά σε θέματα ποινικού δικαίου χρησιμοποιείται αυτό του τύπου το νομικό κείμενο παρόλο που οι κανονισμοί χρησιμοποιούνται πολύ συχνά σε θέματα συνεργασία σε αστικές υποθέσεις ορισμένα κράτη-μέλη επιθυμούν οδηγία αντί για κανονισμό. Τα, η άποψη των κρατών μελών είναι διχασμένη και η Προεδρία θα συνεργαστεί με την Κομισιόν και με τον Κοινοβούλιο για να βρούμε την πιο κατάλληλη λύση. Αυτό θα ε, επιτρέψει, αν τα καταφέρουμε, ε, να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις ε, με το Κοινοβούλιο στην αρχή του 2018. Πρόληψη και διαρεύνηση ε, ποινικών ε, μάλλον εγκλημάτων και πρόσβασης και στα δεδομένα και ανταλλαγή πληροφοριών είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ε, θα πρέπει να βρούμε μια κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα στην ιδιωτικότητα και την ασφάλεια, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τους κανόνες ε, για την διατήρηση στοιχείων ε, τηλεπικοινωνιών. Η ομάδα εργασία για την ανταλλαγή πληροφορίας και την προστασία των δεδομένων, η DAPEX, συνέρχεται στο, με τη μορφή των φίλων της Προεδρίας για να επιτρέψει να γίνουν συζητήσεις για τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και να δουν ποιες θα είναι οι επιπτώσεις τους. Ε, συνεχίζουμε να ψάχνουμε ε, λύσεις ε, για την ποινική δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου στον κυβερνοχώρο και, για την διαρεύνηση κυβερνοεγκλημάτων και εγκλημάτων που περιέχουν ηλεκτρονικά πιστήρια για να τις κάνουμε πιο αποτελεσματικές. Θα δούμε τι τα προβλήματα που δημιουργούνται. Πολύ συχνά τα ηλεκτρονικά πιστήρια βρίσκονται σε άλλες χώρες εκτός των χωρών που γίνεται η έρευνα και γι' αυτό λόγο πρέπει να δούμε πώ μπορούμε να συνεργαστούμε διασυνοριακά. Περιμένουμε την, ε, με ανυπομονησία την πρόταση της Κομισιόν ε, για την, τα ε, ηλεκτρονικά πιστήρια που θα δημοσιευθεί φέτος. Γνωρίζουμε ότι η Κομισιόν αναλύει αυτή τη στιγμή τις τεχνικές και νομικές πτυχές που σχετίζονται με την κρυπτογράφηση και το πώς επηρεάζει η κρυπτογράφηση τι ε, ποινικέ έρευνες. Είναι πολύ σημαντικό θέμα και διχάζει. Ε, πριν βιαστούμε να βρούμε λύσεις θα πρέπει να ε, σταθμίσουμε τα συμφέροντα όλων των φορέων που εμπλέκονται, όλων των εμπλεκομένων και να, τα αναλύσουμε. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες ε, για τα, για ε, τα ποινικά μητρώα ε, και πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολιτών τρίτων ε, χωρών. Γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι θα πρέπει να διευρύνουμε το σύστημα των ευρωπαϊκών ποινικών, σύστημα πληροφοριών ευρωπαϊκών ποινικών μητρώων για να επιτρέψουμε την ανταλλαγή πληροφοριών και για επικόστερη των χωρών. Η Κομισιόν υπέβαλε μια αρχική πρόταση διοδηγία το 2016, αλλά οι διαπραγματεύσει είχαν ανασταλεί γιατί το Συμβούλιο ζήτησε ε, να δημιουργηθεί ένα τέτοιο σύστημα, ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών για επικόστερη των χωρών ω ένα κεντρικό αυτοματοποιημένο σύστημα. Η Κομισιόν υπέβαλε μια πρόσθετη πρόταση πριν από δύο εβδομάδε και το Συμβούλιο θα ξεκινήσει να την εξετάζει το την επόμενη εβδομάδα. Και οι δύο προτάσεις είναι πολύ σημαντικές και σκοπεύουμε να τις συζητήσουμε παράλληλα στο Συμβούλιο. Στόχος μας είναι να φτάσουμε σε μια γενική προσέγγιση και για τις δύο προ... προτάσεις, την οδηγία δηλαδή και τον κανονισμό, μέχρι το τέλος της Εστονικής Προεδρίας. Ένα σημαντικό τμήμα αυτού του συστήματος είναι μια κεντρική ε, βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ε, δακτυλικά αποτυπώματα που θα επιτρέπει ε, την ταυτοποίηση των υπηκών τρίτων χωρών. Τώρα, περνάω στην προστασία των δεδομένων. Ε, Ένα από τους ε, ε λήθου τη ενιαία ψηφιακή αγορά είναι η προστασία των δεδομένων. Τον Ιανουάριο του 2012 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε μια συνολική μεταρρύθμιση του καθεστώτος της προστασίας των δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως γνωρίζετε, το Συμβούλιο θέτησε μια γενική προσέγγιση για τον κανονισμό, για, την προστασία, για τους κανόνες προστασίας των δεδομένων στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Ιούνιο του 2017. Εμείς είμαστε έτοιμοι και πρόθυμοι να διαπραγματευτούμε εκ μέρους του Συμβουλίου μόλις το Ευρωπαϊκό ε, Κοινοβούλιο υιοθετήσει τη θέση του. Είναι σημαντικό επίσης ο κανονισμός να εφαρμοστεί ταυτόχρονα με τον κανονισμό ε, γενικής, με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας των Δεδομένων τον επόμενο Μάιο. Ε, επιπλέον των κανόνων προστασίας των δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δούμε και τη συνολική εικόνα. Ως Προεδρία θα διευκολύνουμε ε, την ε, ένταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πρόσθετο πρωτόκολλο του Συμβουλίου της Ευρώπης, τη Σύμβαση Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των δεδομένων. Είναι η Σύμβαση 108. Η ε, σύναψη αυτής της, αυτού του πρόσθετου πρωτοκόλου θα ε, φέρει πιο κοντά τους δικούς μας κανόνες με, τον, με τους υπόλοιπους ευρωπαϊκούς. Τώρα, ε, θεμελιώδη δικαιώματα. Ο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών και του κράτους δικαίου είναι ακρογωνία ηλίθη των νομικών συστημάτων των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Εστονία θα στηρίξει αυτές τις αρχές κατά τη διάρκεια των ασιών του Συμβουλίου. Στόχος μας είναι να γίνει μια συζήτηση για το κράτος δικαίου στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων. Η αξιολόγηση της εμπειρίας που αποκτήσαμε κατά τη διάρκεια των ε, δύο ετήσιων διαλόγων του Συμβουλίου για το κράτος δικαίου δείχνει την ανάγκη να συνεχίσουμε και να εντείνουμε το διάλογο στο Συμβουλίο. Προς αυτήν την κατεύθυνση κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας θα γίνει ένας ε, διάλογος, μια συζήτηση για την πολυφωνία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το κράτος δικαίου στην ψηφιακή εποχή. Για να προετοιμάσουμε αυτή τη συζήτηση θα διοργανώσουμε ένα σεμινάριο και εκεί καλούμε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πιστεύουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μοιράζονται τις ίδιες απόψεις σε ό,τι αφορά την πολυφωνία των μέσων ε, και την εμπιστοσύνη στα μέσα ενημέρωσης που είναι απολύτως απαραίτητοι όροι ε, για να λειτουργήσει σωστά η δημοκρατία μας προστατεύσουμε και να προωθήσουμε τα θεμέλια δικαιώματα και τι ελευθερίε των Ευρωπαίων πολιτών, θα διασφαλίσουμε τη συνέχεια των δραστηριοτήτων τη ε, ε Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα με την υιοθέτηση απόφαση του Συμβουλίου. Είναι ε, ε για το πολιτέ ε, πρόγραμμα πλαίσιο για την υπηρεσία πριν το τέλο του 2017. δεν είχαν υποστηρίξει πλήρω βέβαια τα κράτη-μέλη το πεδίο εφαρμογή αυτών των δραστηριοτήτων προς το πρότυπο η Κομισιόν. Ε, επίσης, ε, θέλουμε να προωθήσουμε την ε, ε, σύναψη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, της ε, Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης. Ε, επίσης θα γίνει μια συζήτηση για την ετήσια έκθεση της, ε, για την υπηρεσία και την ετήσια έκθεση για την εφαρμογή ε, του, του, της χάρτας των, θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ε, τώρα, πριν από ένα μήνα, στις 8 Ιουνίου, το Συμβούλιο ε, κατέληξε σε μια γενική απόφαση για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Αυτό ήταν αποτέλεσμα σχεδόν τεσσάρων ετών ε, διαπραγματεύσεων με πολλά προβλήματα. Πολλά ζητήματα όπως η ανεξαρτησία του εισαγγελέα, ε, το παραδεκτό των ε, αποδεικτικών στοιχείων κλπ. δημιουργούσαν προβλήματα στα κράτη-μέλη. Όλα αυτά τα θέματα έχουν μακρά ιστορία στα εθνικά δικαιοδοτικά συστήματα και χρειαζόταν βαθιά ανάλυση για να βρεθούν λύσεις. Για αυτόν τον λόγο οι διαπραγματεύσει κράτησαν ε, πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Κάποιοι λένε ότι θα μπορούσε να είναι πιο φιλόδοξο ο κανονισμό. Για τον ίδιο λόγο θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποτελεί πραγματικό επίτευγμα το ότι φτάσαμε σε μια συμφωνία, έστω και σε αυτό το κείμενο. Το κείμενο αυτή τη στιγμή του κανονισμού είναι αποτέλεσμα πολλών συμβιβασμών πράγματι, αλλά το τελικό αποτέλεσμα είναι υψηλή ποιότητα κατά την άποψή μου. Παρ' όλα αυτά, κατέστησα σαφές στην αρχή του χρόνου ότι δεν θα ήταν δυνατόν να εξασφαλίσουμε ομοφωνία. Γι' αυτό το λόγο η ενισχυμένη συνεργασία ξεκίνησε φέτος με 20, με 20 κράτη-μέλη. 20 κράτη-μέλη έχουν ήδη γνωστοποιήσει ότι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ενισχυμένη συνεργασία. Επίτευγμα και αυτό. Πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή και ποια είναι τα επόμενα βήματα. Κατά διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων, από όταν επετεύχθη η γενική προσέγγιση, ε, ελέγχθηκαν οι γλωσσικές εκδοχές του κειμένου από τους γλωσσομαθείς νομικούς. Το κείμενο πέρασε από την Κορεπέ την περασμένη εβδομάδα και το Συμβούλιο θα υιοθετήσει τελική εκδοχή στις 17 Ιουλίου. Μετά από αυτό, το συντομότερο δυνατό θα υποβάλουμε το κείμενο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα ζητήσουμε τη σύμφωνη γνώμη σα, όπω ακριβώ προβλέπει το άρθρο 86 τη Συνθήκη. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα πρέπει να δημιουργηθεί το συντομότερο δυνατό, δηλαδή το 2020 και να αρχίσει να λειτουργεί αμέσω. Ελπίζουμε ότι θα μα δώσετε σχετικά γρήγορα την ε, σύμφωνη γνώμη σα. Το ζητώ αυτό ταπεινά, έτσι ώστε ο οργανισμός να υιοθετηθεί οριστικά τον Οκτώβριο φέτος. Εκ μέρους του Συμβουλίου θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά το Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα τα μέλη της Επιτροπής αυτής για την εξαιρετική συνεργασία που έδειξαν με τις διαδοχικές προεδρίες του Συμβουλίου. Το Συμβούλιο προσπάθησε να πάρει υπόψη της θέσης του Κοινοβουλίου, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την άσκηση των αρμοδιοτήτων ε, και τις ε, ε, σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των κατηγορουμένων. Το Συμβούλιο στο τέλος των διαπραγματεύσεων επίσης είχε και μια καινούργια παράγραφο για το καθεστώς των μη συμμετεχόντων κρατών μελών στο άρθρο 105 μετά από αίτημα του εισηγητή και των συνεισηγητών. Τέλος, να υπογραμμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα είναι αρμόδια και για ορισμένες περιπτώσεις ε, απάτης ΦΠΑ, δεδομένου ότι μετά το αίτημα του Κοινοβουλίου συμπεριλήφθησαν ε, στο πεδίο εφαρμογή. Οπότε ελπίζω ότι εκτιμάτε τις ε, προσπάθειές μας να ικανοποιήσουμε και, το, και εσάς, ε, ιδιαίτερα τις προσπάθειες που έγιναν στο τέλος της Μαλτέζικης Προεδρίας. Ε, θέλουμε πραγματικά, ειλικρινά, να συνεργαστούμε μαζί σας. Ευχαριστώ. Um, Ευχαριστούμε πολύ. Θα περάσουμε πρώτα στους συντονιστές. Ρομπέρτα, είσαι έτοιμη να ξεκινήσεις. Εντάξει, Μπριγκίτ, παρακαλώ. First, um, coordinators first and... Θα ακούσουμε πρώτα τους συντονιστές λοιπόν από τους ε, Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, η Μπριγκίτ Σίπελ. Ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ που είστε ε, εδώ και μα παρουσιάσετε τι προτεραιότητε για την προεδρία σα. Είμαι πεπισμένη ότι θα σημειωθεί κάποια πρόοδο ό,τι αφορά την προστασία δεδομένων. Ξέρετε ότι έχει τεθεί επιτάπητο ε, ιδιωτική σφαίρα και μάλιστα στον κυβερνοχώρο. Ε, θέλουμε να πετύχουμε καλά αποτελέσματα στον τριμερή διάλογο. Ε, Μάριο Λάουστιν, ε, ξέρετε ότι εργάζεται πολύ σκληρά για να έχουμε το ίδιο επίπεδο προστασία όπω και στον κανονισμό Προστασία δεδομένων. Σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είναι καλό που τελικά θα έχουμε τουλάχιστον 20 ε, κράτη-μέλη για αρχή και αυτό είναι ε, μεγάλη επιτυχία μετά τις συζητήσεις που κάναμε τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Παρ' όλα αυτά θέλω να εξετάσω λίγο πιο μακρόπνο αυτό το σχέδιο. Έχετε κάποιες ε, κάποια εικόνα ή θεωρείτε ότι το Συμβούλιο μπορεί να ασχοληθεί περισσότερο με αυτό το ζήτημα για να πείσουμε και άλλα κάτι μέλη να συμμετάσχουν στο σύστημα. Γιατί λυπάμαι που τελικά δεν θα συμμετάσχουν όλα τα μέλη. Ιδίω ε, σε κάποιες χώρες ε, για τις οποίες υπάρχουν εκθέσεις από τον Όλαφ, για παράδειγμα, που καταδεικνύουν ότι θα έπρεπε να συμμετάσχουν. Εκτιμώ ιδιαίτερως τη στήριξή σας ε, προς τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων σε ό,τι αφορά την ε, σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, ε, θα συμφωνήσετε κι εσείς ότι αυτό μπορεί να γίνει όντως ε, κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι κάτι στο οποίο προσβλέπουμε ιδιαίτερως και κάτι τελευταίο. Ή μάλλον όχι. Θα μείνω εδώ. Ευχαριστώ. Και εγώ έτσι <laughs> λέω. Όχι για εσάς βεβαίως, γενικότερα. Ούτε εσείς θέλετε να πάρετε το λόγο. Τι έχετε πάθει σήμερα. Νάταλη. Ναταλή, ξέρω ότι σίγουρα εσύ θα θες να μιλήσεις για τους ε, φιλελευθέρους. Ευχαριστώ, Κλόντε. Ευχαριστώ και τον ε, κύριο Υπουργό που ήρθε στην Επιτροπή μας μερικές μέρες μετά τη συναντησή μας στο Ταλίν. Σας ευχαριστώ λοιπόν που είστε εδώ και για την παρουσίαση που κάνατε για τις προτεραιότητες ε, της Προεδρίας σας μια προεδρία που θα είναι πολύ σημαντική, στρατηγική σημασία για την Ευρώπη, εφόσον για πρώτη φορά αναλαμβάνει την προεδρία ως ε, χώρα. Σας ε, ευχαριστώ για όλα τα σημεία που θίξατε, αλλά και που επιμείνατε σε συγκεκριμένα ζητήματα ε, δικαστικής συνεργασία στο ποινικό δίκαιο, που είναι δύσκολα να εναρμονιστούν, γιατί υπάρχουν διαφορετικές παραδόσεις ε, και κουλτούρες στι επιμέρους χώρες. Όμως αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό για την Ευρώπη, ή τουλάχιστον όπω εμεί επιθυμούμε να δούμε την Ευρώπη. Θα επιμείνω σε ένα σημείο το οποίο θίξατε και εσεί προηγουμένω μετά το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών ΔΕΗ ε, στο Ταλίν. Υπήρχε λοιπόν αυτός ο φάκελος για την καταπολέμηση της ε, τρομοκρατίας και των ε, πηγών χρηματοδότησης τρομοκρατίας και για τον κανονισμό ε, για τα μέτρα της δίμευσης και κατάσχεσης. Είναι εξαιρετικά σημαντικός αυτός ο φάκελος, μεταξύ πολλών άλλων βεβαίως που είναι πολύ σημαντικά για εσάς και για την Επιτροπή μας. Θα ήθελα μόνο να σταθώ στο εξή. Ε, σε ό,τι αφορά την ε, ε, δίμευση των προσόδων από κλιματικέ ενέργειε που ανέρχονται σε δισεκατομμύρια το ευρώ, χρειαζόμαστε ταχύτατη ανάληψη δράση και αντιμετώπιση, γιατί και οι εγκληματίε, όπω ξέρουμε, πολύ συχνά ενεργούν πιο γρήγορα από εμά. Σε ό,τι αφορά τώρα την νομική μορφή που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, για αυτό το εργαλείο που είναι το, το εργαλείο του κανονισμού. Το αναφέρατε κι εσείς. Θα ήθελα ε, να μου πείτε ποια θέση θα λάβει η Προεδρία σας. Φαντάζομαι ότι ως ε, φιλευρωπαϊστές θέλετε ένα ποιοτικό άλμα προς τα μπρος, δηλαδή με την αξιοποίηση ενός κανονισμού και όχι μιας οδηγίας. και κατανόησα την ουσία των όσων είπατε, όμως δεν κατάλαβα τελικά ποια είναι η θέση της Προεδρίας. Εσείς τι θα επιδιώξετε ενώπιον των ομολόγων σας που λίγο ακόμα διστάζουν ε, να υιοθετήσουν έναν κανονισμό που μπορεί να μας ε, δώσει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Ευχαριστούμε Ναταλή. Υπήρξε μια τεράστια συζήτηση για αυτό το θέμα το Συμβούλιο των Υπουργών, όμως νομίζω ότι υπήρχε δικογνωμία μεταξύ των κρατών μελών. Εμείς προφανώς και θέλουμε κανονισμό. Σας ευχαριστώ. Η Ρομπέρτα Μέτσολα από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τον Υπουργό που μας παρουσίασε τις προτεραιότητες της Εστονικής Προεδρίας. Ευχαριστούμε και για όλο το προπαρασκευαστικό έργο που έχετε κάνει στους τελευταίους ε, μήνες ήρθατε σε επαφή μαζί μας, ήρθατε να μας μιλήσατε και, μιλή... ζητήσατε να σας πούμε και τις ε, προτεραιότητες της κάθε πολιτικής ομάδας. Εγώ θα ήθελα να σταθώ στην ε, Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Θα ήθελα τουλάχιστον στο το τέλος της διαδικασίας ε, σύστασης της εισαγγελίας να προσπαθήσετε να διασφαλίσετε ότι θα συμμετάσχουν τελικά όλα τα κράτη-μέλη, συμπεριλαμβανομένου και του δικού μου για να έχουμε όσο γίνεται περισσότερα κράτη-μέλη ε, που θα συμμετάσχουν στην ε, λήψη αυτής της απόφασης για την ε, σύσταση αυτής της αγγελίας, ιδίως ό,τι αφορά τις εγκληματικές ενέργειες και τα έσοδα από τις εγκληματικές ενέργειες. Από την άλλη θέλουμε να υπάρχει κάποιο ψήφισμα ή μάλλον κάποια επίλυση και διέξοδο στις διαπραγματεύσεις για την καταπολέμηση του ξεπλήματος νομικού χρήματος και ελπίζουμε να γίνει αυτό εντός του επόμενου εξαμήνου και να υπάρχει πραγματική επιτυχία στις διαπραγματεύσεις για τις οποίες είστε αρκετά αισιόδοξου με ιδιαίτερο Και η Τζούντιθ Σαργεντίνη για τους Πρασίνους. Just... Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Δύο ζητήματα θα ήθελα να επισημάνω. Αρχικά, να σας συγχαρώ για την ανάληψη των καθηκόντων σας. Βέβαια, όταν μια χώρα αναλαμβάνει δεύτερη, στο δεύτερο εξάμεινο δηλαδή την Προεδρία, βρίσκεται σε μια δύσκολη θέση γιατί έχουμε και τις θερινές διακοπές, ε, μετά τρεις μήνες δουλειά και ξαφνικά φτάσαμε Χριστούγεννα ενώ έχετε πάρα πολλά, πάρα πολλά πράγματα να κάνετε με ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα. Είμαι συνεισηγήτρια στην ε, οδηγία για το ξέπλυμα βρωμικού χρήματο. Δεν έχουμε ολοκληρώσει τι ε, διαπραγματεύσει υπό την Μαλτεζική Προεδρία και μάλιστα θα ξεκινήσουμε αύριο το πρωί ένα νέο τριμερή διάλογο με τους αισθονού συναδέλφους σας. Εκτιμώ ιδιαίτερως ε, τις επαφές που είχαμε ήδη στις προετοιμασίες μας για να διευκρινίσουμε και την εντολή του Συμβουλίου, το Κοινοβούλιο επιθυμεί να ενισχυθεί η διαφάνεια ε, του δικτυωσιακού καθεστώτος και επιχειρήσεων και καταπιστευμάτων. Αυτό σίγουρα αποτέλεσε σημείο ε, εξέτασης ε, και σε ό,τι αφορά τα έγγραφα του Παναμά για την φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή εκτιμούμε ότι η Εστονία ε, φημίζεται για την προσήλωση στη διαφάνεια που έχει. Οπότε προσβλέπω και εγώ στη συνέχεια των διαπραγματεύσεων ε, και στην εξέβρεση ε, σημαντικών λύσεων σε αυτές τις διαπραγματεύσεις το φθινόπωρο. Τώρα, στο πρόγραμμά σας θέλετε να ξεκινήσει και πάλι συζήτηση για την διατήρηση των δεδομένων. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το αναπτύξετε αυτό λίγο περισσότερο. Υπήρξαν κάποιες υποθέσει ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου πριν από μερικά χρόνια και ε, ε, ουσιαστικά ακυρώθηκε η ευρωπαϊκή νομοθεσία σε αυτό το πεδίο. Τα κράτη-μέλη αναγκάστηκαν να αλλάξουν ε, την πολιτική τους τίποτα δεν αντικατέστησε την ε, σχετική νομοθεσία για την διατήρηση δεδομένων. Στο Κοινοβούλιο αμφιβάλλουμε κατά πόσο μπορείτε να καταλήξετε σε νέα νομοθεσία που θα λαμβάνει υπόψη ε, τις επισημάνσεις του δικαστηρίου. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε ε, δύο πράγματα παραπάνω για τα σχέδιά σας ό,τι αφορά την ε, διατήρηση των δεδομένων. Ευχαριστούμε, Τζούντιθ. Συγγνώμη, Μαρτίνα και εσύ ε, θα πάρεις το λόγο εξ ονόματος ε, της ΓΚΟΕ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον Υπουργό για τις προτεραιότητες που μας παρουσίασε, ιδίως ε, για την αναφορά σας στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και στη Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, πιο συγκεκριμένα και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Μιλήσατε και για την απασχόληση και την ασφάλεια. Και επειδή έχουμε και διάφορες ε, ρήτρε opt-in και opt-out ε, στη δικαστική νομοθεσία και επειδή έχουμε και το Brexit ε, το οποίο πλησιάζει, εγώ ήμουν και η συγγήτρια στις ε, ψυχοτρόπες ε, ουσίες, ε, τις νόμιμες όμως ναρκωτικές ουσίες τελικά. Σε κάποιες περιπτώσεις στην Ιρλανδία είχαμε δύο διαφορετικά ρυθμιστικά πρότυπα, ένα για τον νότο και ένα για τον βορρά της νήσου. Και αυτό οδήγησε σε αύξηση του λαθρεμπορίου. Προφανώς και χρειαζόμαστε μια ενιαία προσέγγιση που τελικά βέβαια αυτό θα πληγεί εξαιτία του Brexit, ιδίω αν πρόκειται για ένα σκληρό Brexit, ε, από ό,τι φαίνεται αυτή την άγουσα ακολουθεί η Βρετανική κυβέρνηση. Επειδή έχουμε θάλασσα, έχουμε λιμένες, ε, όλα αυτά είναι ε, μια ανοιχτή επικράτεια και υπάρχουν πολλοί τρόποι παράνομης διακίνησης αυτών των προϊόντων την Ιρλανδία υπάρχουν όμως 197 ε, ε, σημεία συνόρων που ουσιαστικά είναι αδύνατο να κλείσουμε, να στεγανοποιήσουμε τα σύνορα εκτός και αν ε, υψώσουμε ένα τείχος όπως αυτό που θέλει να φτιάξει ο Τραμπ. Δεν ξέρω λοιπόν τι πρόκειται να γίνει δεδομένου και του χρονικού περιορισμού λόγω των θερινών διακοπών και επειδή θα χάσουμε χρόνο έτσι. Κάτι όμως το οποίο ήθελα να αναφέρω για τις επιπλοκές ε, του Brexit και τις προεκτάσεις για την Ιρλανδία. Υπάρχει υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, να ε, διαφυλάξει την Συμφωνία Good Friday σε όλα τα τμήματα. Υπάρχουν και εχέγγυα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μιλήστε εσείς και για τη χάρτα των ανθρώπινων δικαιωμάτων και όλα τα σταγματικά και πολιτικά δικαιώματα και συγκεκριμένα το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης. Και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το οποίο μπίπτει στο δικό σας τομέα αρμοδιοτήτων, είναι αυτό το οποίο επιλαμβάνεται αυτών των υποθέσεων. Για τους επόμενους μήνες πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτή η συμφωνία στην Ιρλανδία ε, και η διαφύλαξη της σε όλα τα τμήματα σημαίνει αυτό ακριβώς. Αυτή είναι και η θέση του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Για να προστατεύσετε όλα τα τμήματα της συμφωνίας, η κυβέρνηση στη Βόρεια Ιρλανδία μπορεί να υιοθετήσει και να θεσπίσει ε, νόμους ε, μόνο αν συμμορφούνται με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Ε, δεν γίνεται να έχουμε δύο λοιπόν διαφορετικά πρότυπα στην ίσο όπως έγινε με τις ψυχοτρόπους ουσίες. Εντός λοιπόν αυτού του εξαμήνου ξέρω ότι θα υπάρξουν και άλλα πράγματα τα οποία ε, θα πρέπει ε, να σας απασχολήσουν, πιο συγκεκριμένα και για το Brexit. Θέλω λοιπόν να το έχετε αυτό κατά νου. Μπορεί να υπάρξει, ε, να ζημιωθεί η μοναδική ειρηνευτική διαδικασία στην οποία εμπλέκεται αυτή τη στιγμή η Ευρώπη. Γι' αυτό πρέπει να δούμε κατά πώς θα παραμείνει και η Βόρεια Ολλανδία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και Κάποιοι λένε ότι θα μπορούσε απευθείας μετά το Brexit να ε, επανενταχθεί η Βόρεια Ολλανδία στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε πολύ Μαρτίνα. Ε, ανέδειξε συνάδελφο ένα από τα βασικά ζητήματα των ε, διαπραγματεύσεων ε, του Brexit, που είναι και το θέμα της Βορειοϊρλανδίας. Είναι κάτι το οποίο σίγουρα θα σα ενδιαφέρει ιδιαίτερω. Ευχαριστούμε τη Μαρτίνα που το έδειξε. Κατερίνα Τσινίτση, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, και σας και καλωσορίζουμε τον Υπουργό στην Επιτροπή μας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ ε, για την παρουσίαση των προτεραιοτήτων κατά αυτό το εξάμενο. Και εγώ, όπως και όλοι οι συνάδελφοι, θέλω να αφαιρθώ σε θέματα τα οποία έχουμε στην καρδιά μας. Παρακολουθούμε βέβαια με μεγάλο ενδιαφέρον τα θέματα της δικαιοσύνης και της ασφάλειας. Εγώ προσωπικά προέρχομαι από την Ιταλία, πιο συγκεκριμένα από τη Σικελία και είμαι δήμαρχος και έχουμε την, ε, την εμπειρία επίσης τη δικαστική ε, Θεωρώ λοιπόν και είμαι πεπισμένη για τη συνεργασία. Συνεργασία η οποία και αυτές είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε αντιμετωπίζουμε εμείς, αλλά προφανώς αντιμετωπίζει και η Ιστονική Προεδρία, ε, μία συνεργασία η οποία περνάει μέσα από τα ηλεκτρονικά συστήματα. Ε, είχα τη δυνατότητα να επισκεφτώ την EU και είμαι και σχεδόν συγγήτρια των Σοσιαλδημοκρατών για τον νέο για το EU Ξέρω λοιπόν πώς λειτουργεί αυτός ο θεσμός και λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Παρ' όλα αυτά χρειαζόμαστε ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο για να ε, μπορεί και η EU να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις. Όπως και χθε, ε, στον Υπουργό Εστερικών. Θέλω να μας πείτε ποια είναι η άλλη πλευρά του νομοθετικού νομίσματος, δηλαδή αποτελεσματική συνεργασία για τα πληροφορικά συστήματα και ε, εκείνο που είναι ιδιαίτερα σημαντικό είναι το θέμα της διαλειτουργικότητας. Θα ήθελα να έχω την άποψή σας και από αυτού, γιατί πιστεύω ότι η διαλειτουργικότητα είναι απαραίτητη για να έχουμε ένα σύστημα πληροφορική το οποίο θα συγκεντρώνει δεδομένα και θα είναι αποτελεσματικό. Για το άλλο θέμα μίλησαν πάρα πολλοί συνάδελφοι. Ε, πρόκειται για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Συμφωνώ μαζί σας ότι θα έπρεπε να έχουμε ε, μια πιο φιλοδοξία ε, εισαγγελία. Ε, εν πάση πτώση, τα 27 από τα 28 κράτη καλό είναι. Και θέλω να ρωτήσω, αναφερόμενοι και σε αυτό που είπε η κυρία Ζίπελ, ε, δηλαδή ε, τι θα κάνετε για να πείστε και τις άλλες χώρες να προσχωρήσουν, γιατί παραμένει ένα πλαίσιο, ένας χώρος που δεν θα καλύπτεται, επειδή δεν θα είναι όλα τα κράτη-μέλη, δεν θα συμμετέχουν όλοι και ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλοί που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν αυτά τα κενά. Σας ερωτώ λοιπόν, λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό, αυτός ο κενός χώρος έχει σχέση και με τη δουλειά που κάνει η Eurojust, θέλω να μας πείτε Όσον αφορά τη Eurojust και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μήπως το Συμβούλιο έχει σκεφτεί πώς θα πρέπει να ρυθμιστούν οι σχέσεις ανάμεσα ε, στους δύο αυτούς φορείς. Ε, μιλήσατε επίσης ε, για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και εδώ θέλω να σας πω ότι αυτά είναι θέματα που είναι βαθιά στην καρδιά μου. Η δίμευση είναι ένα μέτρο το οποίο έχει καταστεί πολύ αποτελεσματικό, αυτό έχουμε τουλάχιστον ε, διαπιστώσει στη χώρα μου. Θέλω λοιπόν να μας πείτε ε, τι ακριβώς πιστεύετε σχετικά με το θέμα αυτό, τι πιστεύει το Συμβούλιο. Και τέλος θα ήθελα να μας ενημερώσετε για το θέμα της δικαιοσύνης, της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης. Γιατί είναι αλήθεια ότι τώρα πια ε, μπορούμε να βασιζόμαστε σε συστήματα πληροφορικής που είναι αρκετά αξιόπιστα όπως το σύστημα της Europol. Δυστυχώς όμως ε, κάτω από την πρόφαση την ε, δικαστική και νομοθετική ρύθμιση έχουμε καθυστερήσει και όσον αφορά και το EU Codex και άλλα συστήματα. Εγώ πιστεύω ότι και αυτά πρέπει να είναι προτεραιότητες, επ' αυτών πρέπει να δουλέψετε έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα οι προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστώ πολύ και θα μιλήσω εστονικά γιατί έχουμε κοινή γλώσσα με τον κύριο Υπουργό. Κύριε Υπουργέ, στην δική σας την ομιλία αναφερθήκατε στο ε, στέσμι μέτρων ε, προστασία δεδομένων. Είπατε ότι τρέχουν παράλληλα πολλές εργασίες. Αυτό βέβαια ε, είναι ένα πολύ σημαντικό πακέτο. Ε, αυτό που είναι, έχει ιδιαίτερη σημασία σε αυτήν την δέσμη μέτρων είναι η ιδιωτική σφαίρα, η προστασία της ιδιωτικής σφαίρας. Εμείς εχθές είχαμε την καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση τροπολογιών. Θα δουλέψουμε επί του θέματος και τα διάρκεια των διακοπών, έτσι ώστε στις αρχές Σεπτεμβρίου να μπορούμε να καταθέσουμε ε, την τελική εκδοχή και να μπορούμε να ψηφίσουμε στην Επιτροπή. Θέλω να ελπίζω ότι η Εστονική Προεδρία ε, θα προχωρήσει κατά τη διάρκεια της Μαλτέζικης Προεδρίας. Δεν υπήρξε πρόοδος. Εσείς ελπίζετε ότι η Εστονική Προεδρία θα προχωρήσει το θέμα της ηλεκτρονικής ε, ε, αλληλογραφίας και προστασίας δεδομένων. Αυτό το θέμα της, των δεδομένων ε, είναι ρεαλιστικό να είναι έτοιμο μέχρι του χρόνου, τον Μάιο. Και έχω και άλλη μια ερώτηση, η οποία αφορά σε ένα πολύ σημαντικό θέμα που είναι ο κανονισμός για την προστασία των δεδομένων ε, που έχει ήδη εγκριθεί. Βλέπουμε υπάρχουν πολλές διαφωνίες όπως και για την οδηγία για την αστυνομία. Αυτά ε, ως Προεδρία θα τα εξετάσετε και τι θα γίνει τελικά όταν θα δεθεί το θέμα της εφαρμογής. Γιατί όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Κανονισμός για την προστασία των δεδομένων ε, μπορείτε κάπως να μας εξηγήσετε πώς ακριβώς παρουσιάζονται αυτά στην ανάλυση σας. Ο κύριος Κώστα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε για όλα αυτά που μας ε, είπατε. Ο κύριος Κώστα. Ε, εδώ και αρκετό καιρό συζητάμε για μια έκθεση πρωτοβουλίας για την ε, προστασία των καταγγελόντων. Από το σκάνδαλο των LuxLeaks υπάρχει εξής κατάσταση. Έχουμε δημοσιογράφους ε, οι οποίοι δίδουν σημαντικές πληροφορίες ε, στην κοινή γνώμη, έχουν σχέση αυτές με την φοροποφυγή, τη φοροδιαφυγή. Τελικά όμως ε, αυτοί οι οποίοι έχουν διαπράξει τη φοροδιαφυγή και φοροποφυγή δεν στυλιτεύονται εκείνοι, αλλά ποιοι στυλιτεύονται οι καταγγέλλοντες. Αυτοί καταλήγουν στα δικαστήρια. Ε, τώρα λοιπόν στο, στο Κοινοβούλιο υπό την Νομική Επιτροπή αλλά και την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ ε, συζητάμε πώς μπορεί να σταματήσει πια αυτό το σκάνδαλο και οι καταγγέλλοντες ε, να χαίρουν ευρεία νομικής προστασίας. Μέχρι τώρα η Κομισιόν έχει πρόβλημα δεν είναι σε θέση να καταθέσει νομοθετική πράξη. Εσείς λοιπόν μπορείτε να φανταστείτε κατά τη διάρκεια της προστασίας σας της Προεδρίας σας, με συγχωρείτε, να βάλετε ως προτεραιότητα το θέμα των, της προστασίας των καταγγελόντων, έτσι ώστε να δρομολογηθεί μια διαδικασία που θα οδηγήσει στην νομική προστασία των καταγγελόντων, των whistleblowers. Σιλβεγγύο, θα είμαι πολύ σύντομη, Πρόεδρε. Γιατί κύριε Τσινίτσι σχολίασε αυτό που ήθελα και εγώ να ρωτήσω. Ε, γίνονται συζητήσεις και έχει ταυτόχρονα μπλοκαριστεί το θέμα της ε, ε, το θέμα του ελέγχου, του συνοριακού ελέγχου. θα ήθελα να θέσω το θέμα της διαλειτουργικότητας γενικότερα σε ό,τι αφορά θέματα εισόδου-εξόδου, αιτίας και λοιπά. Ποια είναι η θέση σας, τι μπορούμε να περιμένουμε. That a short question, but be a long Σύντομη ερώτηση, αλλά θα είναι μακροσκελής η απάντηση, γιατί θίξα το θέμα της διαλειτουργικότητας. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Μπορείτε να ομαδοποιήσετε αν θέλετε. Κατά τη διάρκεια του άτυπου συμβουλίου συναντήθηκα με τον κύριο Μωράης και του είχα εκμυστηρευτεί ότι είμαι λίγο νευρικός. Δεν υπάρχει λόγο να είσαστε νευρικός, να έχετε άγχος. Ε, μου είπε ότι όλα θα πάνε καλά και του είπα το ίδιο λέω και εγώ στην κόρη μου όταν την πάω στον οδοντίατρο. Τουλάχιστον είσαστε ειλικρινείς και μας το λέτε. Ε, ευχαριστώ πολύ για τις απόψεις που εκφράσατε για όλα αυτά τα σοβαρά θέματα. Να σας πω τις δικές μου σκέψεις. Κύριε Τσινίτσι, ρωτήσατε για την ε, ψηφιακή δικαιοσύνη, την ηλεκτρονική δικαιοσύνη. Το συζητήσαμε και στο Άτυπο Συμβούλιο. Κάναμε μια παρουσίαση για το πώ αντιμετωπίζουμε εμείς αυτό το φιλόδοξο σχέδιο της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης στην Ευρώπη. Και δώσαμε ένα παράδειγμα ε, εσθονικό θα έλεγα. Ο στόχος είναι να ε, άρουμε όλα τα πολιτικά εμπόδια έτσι ώστε η ηλεκτρονική δικαιοσύνη να καταστεί πλήρως λειτουργική παντού σε όλη την Ευρώπη. Όμως υπάρχουν δύο προϋποθέτης. Πρώτον, οι ψηφιακέ δυνατότητες των χωρών μελών, των κρατών μελών και δεύτερον, η διαλειτουργικότητα των συστημάτων. Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας, Ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να προχωρήσουμε στο θέμα της υπηρεσίας EU-LISA ε, που θα μας δώσει ε, κάποιες ιδέες για το μέλλον του e-Codex που είναι ένα πειραματικό πρόγραμμα αυτή τη στιγμή για την δημιουργία μιας πλήρως λειτουργικής ε, ηλεκτρονικής δικαιοσύνης στην Ευρώπη. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα θέματα του ποινικού δικαίου. Σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και το αν θα καταφέρουμε να έλξουμε και τα υπόλοιπα επτά κράτη-μέλη. Θα προτιμούσαμε σίγουρα ως Προεδρία και ως Εστονία αντί για την ενισχυμένη συνεργασία να έχουμε όλα τα κράτη-μέλη με ομοφωνία στο project αυτό. Πρέπει όμως να δεχτούμε την πραγματικότητα. Θα καλωσορίζαμε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος θέλει να συμμετάσχει. Δεν πρόκειται η Ευρωπαϊκή Αγγελία να κλείσει τις πόρτες της. Σε όλες τις περιπτώσεις διαδικασίας ε, ενισχυμένης συνεργασία, πάντοτε τα υπόλοιπα κράτη-μέλη έχουν το δικαίωμα να ε, ενταχθούν στις ενισχυμένε συνεργασίε αργότερα. Και, το ίδιο θα, και αυτό θα κάνουμε και εμείς ως Προεδρία. Θα ενθαρρύνουμε τις υπόλοιπε χώρε που δεν υπέγραψαν την αρχική συνεργασία να το κάνουν. Μερικές φορές βέβαια αυτά τα κείμενα είναι σαν το λαβύρινθο και δεν θα επιθυμούσαν να ξανανοίγαμε, να ξαναξεκινούσαμε τις διαπραγματεύσεις που έχουν ήδη κλείσει. Γιατί κάτι τέτοιο θα μπορούσε να οδηγήσει θάνατο την ε, ενισχυμένη συνεργασία. Ένα άλλο ζήτημα αφορά την διατήρηση των δεδομένων για τις τηλεπικοινωνίες. Πώς θα προχωρήσουμε το ζήτημα. Και αυτό συζητήθηκε με τους Υπουργούς Εσωτερικών στο Τάλιν, στο Άτυπο Συμβούλιο. Η ιδέα που κυκλοφορεί και συζητήθηκε και στο Τάλιν ήταν να συνδεθεί το θέμα αυτό με τον κανονισμό της ε, ηλεκτρονικής ιδιωτικότητας, του e-privacy. Δηλαδή να βρούμε μια ευρωπαϊκή λύση για ε, την διατήρηση των δεδομένων σε συμφωνία με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Το θέμα είναι πολύ ευαίσθητο. Δεν θα πρέπει να βλάψουμε τον κανονισμό για την ηλεκτρονική ιδιωτικότητα κατά τη διάρκεια του άτυπου συμβουλίου. Ήταν σαφές το μήνυμα ότι τα κράτη-μέλη ε, υποστηρίζουν την ανάγκη ε, μιας ε, ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για τη διατήρηση δεδομένων. Όλες, ό,τι όμως και να προταθεί, θα πρέπει να είναι να συνάδει με την φιλοσοφία ε, των αποφάσεων ε, του, Ευρωπαϊκού, του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όπως είπα και στην παρουσίασή μου, συμφωνήσαμε να ζητήσουμε από, την, από μια ομάδα εργασίας να φέρει στο τραπέζι συγγνώμη, να βγάλει από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων ιδέε οι οποίες δεν έχουν λειτουργήσει στο παρελθόν. Θα θέλαμε η Κομισιόν να είναι η υπεύθυνη για την διαμόρφωση αυτής της πρωτοβουλίας, αλλά θέλουμε να του δώσουμε κάποια εργαλεία. Ως, ε, αυτή η Επιτροπή λοιπόν, ως φίλη της Προεδρίας, ε, ε, έχει ως στόχο να υποβάλει διάφορες αναλλακτικές λύσεις. Και στο τέλος του χρόνου θέλουμε να έχει ολοκληρώσει την εργασία της, έτσι ώστε η Κομισιόν να πάρει μια ψυχολογική υποστήριξη, ας πούμε, από την ομάδα εργασίας, για να προχωρήσει γιατί ξέρουμε ότι ως τώρα επικρατεί μια μεγάλη ασάφεια ε, και η Κομισιόν είναι Για την ποινική δικαιοσύνη υπάρχει επίσης και το ζήτημα του πώς μπορούμε να προχωρήσουμε το θέμα των κατασχέσεων και των δεσμεύσεων για ε, αυτή την πρωτοβουλία και το κατά πόσον η Εστονία θα στηρίξει την ιδέα του κανονισμού σε αντιδιαστολή με την οδηγία. Τα κράτη-μέλη είναι διχασμένα μισά-μισά. Σαν τον ε, Ιαννό, μισός-μισός. Ο πρόεδρος λέει, σημειώνω όλες τις εικόνες τις οποίες έχετε χρησιμοποιήσει με το λαβύρινθο, το μηνόταυρο, όλα αυτά. Ε, πολύ γλαφυρή η ομιλία σας. Ε, ο κ. Ρέινσαλου. Εμείς στην Εστονία θέλουμε να βλέπουμε αποτέλεσμα. Άλλο ο στόχος, ο θεωρητικός στόχος. Ασφαλώς και θα προτιμούσαμε έναν κανονισμό. Είναι πιο ισχυρό νομικό μέσον για να επιληθεί το πρόβλημα αυτό. Όμως, αν η μόνη ρεαλιστική επιλογή είναι μια οδηγία, θα την ακολουθήσουμε. Καλέσαμε την Κομισιόν να σκεφτεί καλύτερα ποια είναι η πιο πρακτική λύση για να προχωρήσουμε. Η τελευταία μελέτη της Europol ήταν εντυπωσιακή. Σήμερα 1,1% ε, του κύκλου εργασιών των ποινικών δραστηριοτήτων ε, μόνο ανακτάται. Ο ποινικό δραστηριότητα εννοώ να, ναρκωτικά, οργανωμένο έγκλημα κλπ. Είναι πολύ λίγο. 1,1% του κύκλου ε, εργασιών, των παράνομων αυτών εσόδων από ποινικέ δραστηριότητε ανακτάται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι πρέπει να κάνουμε λοιπόν. Η κυρία Ματίνα αναφέρθηκε στα, στις πτυχές ασφάλειας, η ε, κυρία Μαρτίνα είναι ο μιλητής, ε, στα θέματα στοιχεία ασφάλειας σε ό,τι αφορά τι διαπραγματεύσει με τον Brexit. Και το ζήτημα του λαθρεμπορίου ναρκωτικών. Κατά τη διάρκεια του άτυπου συμβουλίου ε, συναντήθηκα ιδιαίτερος με τον ε, υπουργό δικαιοσύνη, το νέο υπουργό είναι στον κύριο Λίβινγκτον. Έχω και το κινητό του εδώ, για να συζητήσουμε σοβαρά θέματα. Η άποψη τη προεδρία είναι ότι αν θέλουμε η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι ισχυρή στις διαπραγματεύσεις και το αποτέλεσμα να είναι θετικό, ιδιαίτερα για τους πολίτες μας, τότε η... την εντολή διαπραγμάτευσης πρέπει να την εκτελέσουν αυτοί οι οποίοι το έχουν αναλάβει. Αυτοί στους οποίους έχει ανατεθεί η εντολή. Το σημαντικό πάντως είναι τα δικαιώματα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η τα θέματα ασφάλεια και εσωτερικών υποθέσεων όμως θα πρέπει οπωσδήποτε να συζητηθούν κατάλληλα κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Πολύ σημαντικό επίσης ήταν και το ζήτημα της ε, ηλεκτρονικής ιδιωτικότητας. Ε, όπως είπε ο, και ο συνάδελφός μου των ιστορικών υποθέσεων είναι προτεραιότητά μας. Γνωρίζουμε το, την ημερομηνία εφαρμογής προτείνει η Κομισιόν. Θα λάβουμε, θα τη λάβουμε υπόψη κατά τον προγραμματισμό των συζητήσεων στο Συμβούλιο. Αλλά, πάντα υπάρχει ένα αλλά. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι η πρόταση καλύπτει μερικά περίπλοκα ζητήματα και επιπλέον έχει πάρει τη μορφή του κανονισμού, άμεσα εφαρμοστέο δηλαδή. Κάτι που θα χρειαστεί, θα αναγκάσει μάλλον τους συνομοθέτες να το εξετάσουν πάρα πολύ προσεκτικά. Θα πρέπει να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα, σαφέστατα, γιατί αν καθυστερήσουμε το καραβάνι θα χάσει τον ορίζοντα. Επίσης θα πρέπει να προχωρήσουμε παράλληλα σε, όλη, σε όλα τα κείμενα της ομάδας αυτής της πρωτοβουλίας. θέμα που εθιγήταν η, το κατά πόσον η Προεδρία θα εξετάσει, θα καλέσει τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν ε, κομμάτια της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων. Η προστασία των δεδομένων είναι σοβαρό ζήτημα. Γνωρίζουμε ότι τα εθνικά ε, συστήματα διαφέρουν πολύ μεταξύ τους. Και εδώ ερχόμαστε στον πυρήνα της πρωτοβουλίας για την καλύτερη νομοθεσία. θα πρέπει να δούμε και εκ των υστέρων ποια είναι η πραγματικότητα. Ε, θα συμφωνήσω μαζί σας λοιπόν. Εμείς κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας ε, έχουμε λάβει υπόψη ε, στις ομάδες εργασίας μας ε, τις, ε, ε τις επιταγές της καλύτερης νομοθεσίας και έχουμε εκδώσει και, μια, και ένα κατάλογο με κατευθύνσεις γραμμέ στους προεδρεύοντες των συνεδριάσεων έτσι ώστε να λαμβάνουν υπόψη τις τεχνικές και τις πρακτικές που επιβάλλονται ε, από ε, την, ε, την ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας της νομοθεσίας. Πάντως ναι, πράγματι χρειαζόμαστε καινούργια νομοθεσία για αυτό το ζήτημα και ελπίζουμε να πάρει τη σκητάλη και η Βουλγαρική Προεδρία. Και μέσω αυτή θα υποστηριχτεί και η πρωτοβουλία της Κομισιόν για καλύτερη ε, νομοθεσία. Ο ε, κ. Κώστρο και η κυρία Γκυγιόμ ε, θίγει το θέμα των whistleblowers, συζητήθηκε και επί Μαλτέζικης Προεδρίας. Στο άτυπο συμβούλιο, όπου τα κράτη-μέλη εξέφρασαν τις απόψεις τους. για το θέμα των καταγγελόντων. Οι απόψεις που εκφράστηκαν βέβαια διέφεραν πολύ μεταξύ τους. Προφανώς όλοι αντιλαμβάνονται ότι αυτό αποτελεί πρόβλημα, αλλά το κατά πόσον θα αντιμετωπιστεί σε εθνικό ή σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι άλλο θέμα. Δεν συμφωνούν τα κράτη-μέλη μεταξύ τους γι' αυτό. Η Επιτρόπος Γιουρόβα κατέγραψε τις ιδέες των κρατών μελών, τις απόψεις τους και θα τις μελετήσει. Ελπίζω. Ε, και μια διαβούλευση από πλευράς κομισιών για αυτό το θέμα. Ε, σε αυτή τη διαβούλευση συμμετείχαν και πολλά κράτη-μέλη. Ε, και η Κομισιόν θα τα λάβει όλα αυτά υπόψη. Αυτή άλλωστε ε, έχει το δικαίωμα ανάλυση πρωτοβουλία. Τώρα το θέμα τη διαλειτουργικότητα. Από το φθινόπωρο η Προεδρία είναι έτοιμη να συνεργαστεί και με εσάς και με την Κομισιόν για να προετοιμάσουμε το έδαφο για τι επερχόμενε προτάσεις για τη διαλειτουργικότητα. Ο στόχος είναι να εξαλειφθούν τα τεχνικά εμπόδια στα δεδομένα, τα οποία ήδη συλλέγονται, έτσι ώστε να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν ακόμα περισσότερο. Βέβαια θα χρειαστεί να συλλέγουμε όλο και περισσότερα στοιχεία και δεδομένα. Οπότε η διαλειτουργικότητα γίνεται ιδιαίτερα σημαντική. Για τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, που επίσης να πω το εξή. Η Προεδρία επιθυμεί μια ολιστική προσέγγιση της εφαρμογής της σύμβασης της Κωνσταντινούπολης. Και χωρίς καθυστερήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. για τις ερωτήσεις σας, για τα σχόλιά σας. Θα είμαστε πολύ συνεργάσιμοι. Φεύγουν κάποιοι συνάδελφοι. Δεν ξέρω κάποιον από αυτούς που μένουν έχουν ε, πάει ποτέ στην Εστονία, όμως ε, θα συμφωνήσουν σίγουρα μαζί μου ότι η αστυνομική πλευρά έκανε μια πολύ καλή αρχή στην Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ιδίω στον τομέα τη δικαιοσύνη. Βλέπω ότι και ο Μάριο είναι εδώ. Η Μαριόν, συγγνώμη. Ξέρει ότι ε, η Εσθονία ηγείται στα ζητήματα ηλεκτρονικής δικαιοσύνης ε, σε όλες αυτές τις πλατφόρμες, ε, παρότι είναι μια μικρή χώρα, υπάρχει λίγο προστιμένη αξία. Κατά τη διάρκεια του άτυπου συμβουλίου, ΔΕΗ, βέβαια, ε, κυριάρχησαν τα πλέγοντα ζητήματα όπως αυτά της Λιβύης. Όμως ε, η Εστονία παρουσίασε και μια πολύ ε, σωστή σειρά προτεραιοτήτων που θα μας απασχολήσουν σίγουρα πολύ. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ και για το χρόνο που μας αφιερώσατε για να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. Για την κυρία Άντερσον τώρα, το ερώτημά σας κυρίως ήταν, αφορούσε το θέμα της ε, στάσης της Βρετανικής κυβέρνησης στις διαπραγματεύσεις και πώς αυτό μπορεί να πλήξει την συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής. Ίσως θα μπορούσε η κυρία Άντερσον γραπτός να τα στείλει, γιατί ξέρω ότι κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σίγουρα θα ανακύψει και πάλι το ζήτημα. Αν μπορεί λοιπόν να μας το στείλει γραπτός, ε, για να μην ε, αμεληθούν αυτά τα ζητήματα. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι και εσάς και την ομάδα σας. Τελικά δεν ήταν και τόσο άσχημα. Ναι, με τη βοήθειά σας ε, πραγματικά επιβίωσα. Σας ευχαριστώ, ειλικρινά. Εφόσον είναι και τελευταία εβδομάδα και για σας πριν από τις τερινές διακοπές, καλό καλοκαίρι σε όλους να ευχηθώ. Ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε μετά το καλοκαίρι. Κυρία Μάκοβα, θέλετε να πείτε κάτι. Μόνικα Μάκοβα, ονομάζομαι από τη Ρουμανία. Θα ήθελα να σας χαρώ για την προεδρία σας. Είπατε ότι είστε μια μικρή χώρα, ναι, αλλά με τα ανώτερα επίπεδα ε, δικαιωμάτων η της δημοκρατίας και το καθεξής στην Ευρώπη. Συγχαρητήρια λοιπόν. Ε, περιμένουμε πολλά από την Προεδρία σας. Ένα ερώτημα. Όπως ε, και πολλοί άλλοι, και εγώ θα ασχοληθώ με το ζήτημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητε που θα ξεκινήσετε υπό την Προεδρία σας. Ε, ήθελα να ρωτήσω αν είναι προτεραιότητα. Ε, ουσιαστικά είχαμε ολοκληρώσει, αλλά έτσι πάντα αυτά στην Επιτροπή Λίμπε. Μπορείτε να απαντήσετε λοιπόν και σε αυτό. Μάλιστα, λέει ο Υπουργό. Ε, με τα χαρά μπορώ να απαντήσω καταφατικά. Είστε έτοιμος για όλα, βλέπω. Ωραία. Σας ευχαριστούμε όλους. Και είτε το πιστεύετε είτε όχι, το επόμενο θέμα που θα μας προσχολήσει είναι καταγγέλλοντες, ακριβώς. Okay, colleagues, let's um, uh, late now, so... Συνάδελφοι, έχουμε καθυστερήσει λίγο. α περάσουμε λοιπόν ε, απευθείας στην έκθεση Μάκη Παντακβετούρα. Ε, για τους καταγγέλλοντες έχουμε 76 τροπολογίες για το σχέδιο γνωμοδότησης. Θα δώσω λοιπόν ε, το λόγο στη Μάιτε. μας παρουσιάσει την γνωμοδότησή της. Bueno, mm, voy a ir muy breve porque vamos con retraso. Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομη γιατί περνάει και η ώρα. Θα ήθελα να τονίσω και πάλι πόσο σημαντικό είναι να, έχουμε ένα ε, πλαίσιο ε, προστασίας των καταγγελόντων. Ε, με τις συστάσεις που υιοθετήθηκαν γνωρίζουμε την σημασία των καταγγελόντων και τονίζουμε ότι θα πρέπει να ε, προστατεύονται οι καταγγέλλοντες. Γι' αυτό είναι προς όφελος ε, του, της, υπηρεσίας που παρέχουν οι καταγγέλλοντες προς ε, το γενικό συμφέρον. Σας ευχαριστώ συνάδελφοι για τις τροπολογίες σας, 76 τον αριθμό. Θα προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε συμβαστικές τροπολογίες τώρα που είμαστε τελική ευθεία. Πάντα ε, δίνοντας έμφαση στα ζητήματα που απασχολούν την Επιτροπή μας. Σημαντικές όλες ε, οι τροπολογίες θα προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε ένα κείμενο το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τις επιθυμίες όλων των πολιτικών ομάδων στο βαθμό που αυτό είναι δυνατόν. Τη 7 Σεπτεμβρίου θα ψηφιστεί η νομοδότηση, θα περιμένω τι παρατηρήσει σα, τη συμβολή σα. Θα σας ευχαριστώ. Um, Ευχαριστούμε πολύ, Μάιτε. Μίραρ και Κώστερ, παρακαλώ. Κύριος Σκέστερ, παρακαλώ. Ah, I'll just take Mr. and let Mr. Mello settle Please go ahead. Thank you, Chair. Dear colleagues. Uh, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση, την υποβολή τροπολογιών μέχρι τώρα. Η εισηγήτρια, κύριε την ευχαριστώ οι 76 τροπολογίε δείχνουν ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για αυτό το θέμα και εγώ, ω εισηγητή συγχρονόματο των ε, Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, ε, μπορώ να πω ότι ένα είναι σημαντικό το θέμα. Ε, Καταγγέλλοντα στο πλαίσιο των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η προστασία των καταγγελόντων είναι κρίσιμη σημασία για, για τον πλουραλισμό, την ελευθεροτυπία, τη δημοκρατία και την ελευθερία. Αφενό έχουμε το θέμα των θεμελιωδών δικαιωμάτων, το οποίο συνδέεται με τους ε, πολίτε, που πρέπει να γνωρίζουν ε, τις ε, παραβιάσεις που σημειώνονται σε αυτό το τομέα. Και αφετέρου, όσοι καταγγέλλονται κακό κείμενα, διαδραματίζουν έναν κρίσιμο ρόλο γιατί αποκαλύπτουν παραβάσεις και παραβιάσεις και την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σε μία από τι τροπολογίε μου, ε, μάλιστα προτείνω να απονέμουμε ένα ευρωπαϊκό βραβείο καταγγελόντων για να αναδεικνύουμε ακριβώς ε, την αξία αυτής της πρακτικής για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και θα ήθελα να ε, αναδείξω το γεγονός ότι αυτή η πρακτική είναι μια μορφή καλής πολιτικής διαγωγής αν θέλετε. σε ό,τι αφορά τις παραβιάσεις ε, που αποκαλύπτονται από τους καταγγέλλοντες, δεν θα πρέπει ε, να αποκαλύπτονται μόνο ε, αδικήματα, ποινικά αδικήματα, αλλά και ε, κακοδιαχείριση, σοφαρές ε, παραβιάσεις άλλου τύπου θα πρέπει να προστατεύονται υπό αυτό το πλαίσιο. Και για να πάμε ακόμα ένα βε, βήμα μακρύτερα, Μπορούμε να μιλήσουμε και για νομοθεσία ε, για τους καταγγέλλοντες. Προτείνω λοιπόν σε τελεγική σκέψη η προστασία των καταγγελόντων να μην περιορίζεται μόνο σε ευρωπαϊκές ε, υποθέσεις και περιπτώσεις, αλλά και σε διεθνείς υποθέσεις. Τουλάχιστον υπάρχει μια ξεκάθαρη, ξεκάθαρη λύση για τους καταγγέλλοντες που εργάζονται ε, σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, αλλά εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης καμία σχέση εργοδότη-εργαζομένου δεν θα πρέπει να περιορίζει την ελευθερία έκφρασης κάποιου. Και κανείς δεν θα πρέπει να την χάνει, να αποτελεί κείμενο αρνητική διάκριση γιατί ασκεί αυτό το δικαίωμα. Πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα ενστάσεων το οποίο να το διαχειρίζεται ε, μια ανεξάρτητη κεντρική αρχή. Έχω ε, προτείνει να συσταθεί ένας ευρωπαϊκός οργανισμός ε, με έδρα, πόρους, ε, προσωπικό ε, και κατάλληλους εμπειρογνώμονες. Θα πρέπει λοιπόν να θεσπιστεί για να βοηθήσει τους καταγγέλλοντες εντός και εκτός Ευρώπης να παρέχει τις κατάλληλες διόδους για να αποκαλύπτουν αυτά τα κακοσκήμενα και να παρέχει συμβουλές. Θα ήθελα επίση να πω ότι οι είναι εξαιρετικά ευάλωτοι ε, σε αντίπεινα και ενεργούν με υψηλό προσωπικό και επαγγελματικό ρίσκο και πολλές φορές πληρώνουν βαρύ τίμημα. Γι' αυτό και θεωρώ ότι μέτρα ελάφρυνσης αυτού του κόστους αλλά και επιπρόσθετη αποζημίωση θα πρέπει να προβλέπετε. Τέλος, θα πρέπει πάνω απ' όλα να ορίσουμε τους καταγγέλλοντες. Από αυτό εξαρτάται και η νομοθεσία. Γι' αυτό αναδεικνύω την ανάγκη ύπαρξης ανεξάρτητου και κοινού ορισμού των καταγγελόντων για να διασφαλίζουμε την κατάλληλη προστασία. Κάθε άτομο το οποίο λοιπόν αποκαλύπτει κάποια παράβαση έχει το δικαίωμα της ένομης προστασίας. Εγώ ως εισηγητής θεωρώ, μάλλον ε, θεωρώ ότι η πρώτη εισηγήτρια είναι μια πολύ καλή βάση. Ε, και θέλω να συνεχίσουμε αυτή τη συνεργασία. Ελπίζω να καταλήξουμε σε ε, ικανοποιητικές λύσεις για μια ισχυρή ε, νομική προστασία των καταγγελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Thank you very much, Mr. Coster. Um, and the EPP shadows, Mr. Mello, please. Ο κύριος Μέλο από το ΕΛΚ. Bom, uh, muito obrigado. Enfim, eu não ia nesta fase de ser muitas considerações. Θα ήθελα να πω ότι κατά την άποψή μου η πρόταση είναι πολύ καλή. Έχω βέβαια κάποιες επιφυλάξεις. Προσπάθησα αυτές τις επιφυλάξεις μου να τις ε, συμπεριλάβω στις ε, τροπολογίες που κατέθεσα και ελπίζω να τα έχετε όλα αυτά κατά νου. Προφανώς λοιπόν έχουμε να κάνουμε με τους ε, καταγγέλλοντες οι οποίοι ε, και αυτοί πρέπει να στηρίζονται σε γεγονότα ή ε, σε πράγματα που γνωρίζουν πολύ καλά. Γι' αυτό λοιπόν οι καταγγέλλοντες πρέπει να προστατεύονται. Ας το δούμε λιγάκι το θέμα από νομική σκοπιά. Ο νόμος ε, μερικές φορές είναι αφηρημένο, είναι γενική, γενικός, πολύ ασαφής. Και μην ξεχνάμε ότι πολλοί εκμεταλλεύονται αυτή την ασάφεια για δικούς τους ε, εγκληματικούς λόγους. Εγώ πρέπει να σας πω ότι έχω κάποιες επιφυλάξεις ε, στο να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο που να ισχύει σε όλα τα κράτη-μέλη. Θα προτιμούσα να ισχύει περισσότερο η αρχή της επικουρικότητας ε, λόγω του ότι υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο για μας ε, να έχουμε ένα ευρύτερο νομικό πλαίσιο αλλά βέβαια θα πρέπει πάντα να δεχόμαστε και να σεβόμαστε την αρχή της επικουρικότητας. Υπάρχει και κάτι στην έκθεση που χάνεται κατά την άποψή μου και προτείνω ως εκ τούτου το εξής. Έχουμε δύο κατηγορίες ατόμων, προσώπων κάποιοι οποίοι έχουν γνώση κάποιων δεδομένων ε, κάποιες πραγματικότητες η οποία μπορεί να ενδιαφέρει τη δικαιοσύνη αλλά δεν έχουν άμεση ε, συμμετοχή αλλά έχουμε και πολλούς άλλους που είναι τα άτομα που έμεσα ή άμεσα ε, συμμετείχαν σε μια παράνομη δραστηριότητα. Και ίσως χρειάζονται διαφορετική αντιμετώπιση. Στο πορτογαλικό δίκαιο ε, γίνεται αυτή η διάκριση. Ε, υπάρχει ε, το plea bargaining στα, στο αγγλοσαξονικό δίκαιο, ε, το οποίο ε, έχει κάνει διάκριση ανάμεσα σε αυτούς που έχουν συμμετοχή σε ένα δίκημα και σε αυτούς που ε, δεν έχουν. Στο ευρωπαϊκό δίκαιο γενικά αν εμπλέκεσαι σε μια ε, περίπτωση αδικήματο και συνεργαστής σου επιφυλάσσει το δίκαιο, η δικαιοσύνη μια πιο ευνοϊκή μεταχείριση. Θα πρέπει να κάνουμε όμω αυτή τη διάκριση. Αν κάποιος εμπλέκεται στην διάπρεξη ενό μιας εγκληματική πράξης, θα πρέπει να έχει ε, μια ευνοϊκή μεταχείριση, για παράδειγμα διαχωρίζοντας τη δική του υπόθεση από την υπόθεση από τις υποθέσεις των υπολείπων κατηγορουμένων. Δεν λέω ότι αυτό είναι μια λύση, λέω ότι είναι μια πρόταση. Έτσι. Ίσως θα μπορούσε να συμπεριληφθεί και αυτή. Ε, αν δεν επιφυλάσσουμε μια πιο ευνοϊκή μεταχείριση σε αυτούς τους ανθρώπους, τότε δεν θα τους δώσουμε κίνητρο. Απ' την άλλη μεριά δεν είναι δυνατόν να εξισώσουμε αυτούς που διέπραξαν ένα έγκλημα, ακόμα και αν συνεργάζονται με τη δικαιοσύνη, με αυτούς που δεν έχουν καμία εμπλοκή. Εντάξει, αυτό δεν έχει ληφθεί καθόλου υπόψη στην πρόταση. Ευχαριστώ. Okay, are you finished? Okay. Okay, right. <laughs> Um, e Η κυρία εκ μέρους της, ε, των ECR, της ομάδας ECR. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να απαντήσω στο συνάδελφό μου, γιατί από αυτού του θέματος εγώ έχω τελείως διαφορετική άποψη και εξάλλου γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ για να συζητήσουμε. Το θέμα, ε, ο αγώνας κατά της ε, διαφθοράς, ε, ε, της νομιμοποίησης των παράνομων εσόδων, αυτό θεωρείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα θέμα που έχει σχέση με την εσωτερική τάξη πραγμάτων στην Ένωση. Και αυτό δεν μπορεί κανείς αφενός να θέλει να το καταπολεμήσει και αφετέρου να προστατεύει τα χρήματα των πολιτών αλλά και την εσωτερική τάξη ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να καταφεύγει στους καταγγέλλοντες. Οποιοδήποτε κράτος επιθυμεί να ε, αποκαλύψει το τι συνέβη, τα κακό σκήμενα, με μεγάλη του χαρά ε, θα χρησιμοποιούσε καταγγέλλοντες, γιατί αυτός είναι και ο ευκολότερος τρόπος ε, να μπορέσει ένας ε, θεσμός ε, να αποκαλύψει τι συμβαίνει. Γι' αυτό και υπάρχει προστασία. Αλλιώ θα χάσουν τη δουλειά του. Οι άνθρωποι αυτοί θα φοβούνται για θέματα παρενόχληση. Παραδείγματο χάρη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσοι θέλησαν να εφαρμόσουν τι οδηγίε Ευρωπαϊκή Ένωση για την προστασία των καταγγελόντων, οι καταγγέλλοντες αυτοί αναγκάστηκαν να φύγουν, η ζωή τους ήταν άθλια, αναγκάστηκαν να πάρουν αναρωτική άδεια ή τους χαρακτήρισαν τρελούς ή ε, τους ε, από τη μία υπηρεσία στην άλλη. Στο τέλος ε, ξαναγκάστηκαν να φύγουν. Αυτοί οι οποίοι είναι στη φυλακή και καταγγείλουν, καταγγέλουν άλλους, αυτοί δεν είναι αυτό που λέμε εμείς ε, whistleblowers. Ε, αυτοί καταγγέλουν κάποιους ε, για να μειωθεί η ποινή τους. Αυτοί όμως για τους οποίους μιλάμε εμείς δεν έχουν καμία σχέση με το ποινικό δίκαιο. Δεν έχουν υποστεί καμία ποινή. Ας πούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάνουν τη δουλειά τους, αλλά δεν τους αρέσει η παραβίαση του δικαίου και τα κακό σκήμενα και γι' αυτό θέλουν να τα καταγγείλουν αυτά και θέλουν να βελτιωθεί η κατάσταση. Μερικοί εξημών συνεργαστήκαμε και δουλεύουμε με καταγγέλντες. Οι άνθρωποι αυτοί αυτό κάνουν. Δεν είναι ανήθικο αυτό που κάνουν. Κάθε άλλο. Εγώ θεωρώ ότι είναι απόλυτα ηθικό σε αυτό αυτό το κοινοβούλιο ή σε άλλους θεσμούς ε, να αποκαλύπτουν κακό κείμενα και να αναλαμβάνουν οι αρχές να τα διαλευκάνουν. Αυτό σας είπα διαφέρει από αυτούς που βρίσκονται στις φυλακές. Δεν είναι αυτή η περίπτωση των καταγγελόντων που συζητάμε εμείς. Εγώ λοιπόν στηρίζω την έκθεση. Έχω συντάξει τροπολογίες για να συμπληρώσω την έκθεση και επίσης θέλω να γίνεται και αναφορά και στη διερευνητική δημοσιογραφία που και αυτή είναι πολύ σημαντική για τις έρευνες που γίνονται για τα οξέπλημα, για καταχρήσεις. Ας πούμε παράδειγμα Panama Papers, για δέστε τι έγινε, πώς αποκαλύφθηκαν. Και αν δείτε και την έκθεση της Επιτροπής του Παναμά θα δείτε πόσο καθοριστική σημασία είναι ο ρόλος των καταγγελόντων, των whistleblowers. Ήθελα και εγώ να έχω πει την άποψή μου επί του θέματος. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Ντένις εκ μέρους της ε, Γκούε παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ Κλόντ. Εγώ νομίζω, καταρχήν, σε επίπεδο στρατηγικής, ακούσαμε την Εστονική Προεδρία να λέγει προβλήματα που υπάρχουν ε, στο Συμβούλιο. Κατά κάποιον τρόπο αυτό το περιμέναμε γιατί αρκετά κράτη-μέλη είπαν ότι υπάρχουν προβλήματα επικουρικότητας. Ε, εν ώψη αυτών, εγώ διαρωτώ με κατά πόσον είναι καλύτερα να ζητήσουμε ένα ευρύτερο εργαλείο ή αν θέλετε ένα συγκεκριμένο τομεακό εργαλείο. Κυρίω και πάλι όταν πρόκειται για οικονομικά συμφέροντα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ω κράτο μέλο, δεν μπορεί κανεί ε, να αρνηθεί ότι όταν πρόκειται για οικονομικά θέματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι πρέπει κανεί να το διαλευκάνει και εδώ δεν τίθεται θέμα επικουρικότητα. και εγώ και η ομάδα μου είμαστε υπέρ του να υπάρχει ένα περιεκτικό ευρύτερο εργαλείο και σε αυτή τη φάση ίσω θα ήταν καλύτερα ε, να προχωρήσουμε όσο μπορούμε ω κοινοβούλιο. Εγώ Είμαι και εισηγητή για τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ελέγχου Προπλογισμών επί του θέματος. Έχουμε λοιπόν μια συζήτηση ε, που λέει είτε να πάμε κατά μέτωπο είτε παράλληλα ε, να έχουμε κατά νου ότι ενδεχομένως να πρέπει να υπάρξει ένα ε, μεταβατικό μέσο ή μια τομεακή προσέγγιση. Αυτά γενικότερα ως στρατηγική. Τώρα για τις τροπολογίες Νομίζω ότι δεν πρέπει να πάμε πιο πέρα από αυτό που ενέκρινε εφέτος το Κοινοβούλιο με βάση μια έκθεση ε, που ε, έχω καταρτήσει για τους καταγγέλλοντες. Το ψήφισμα αυτό υιοθετήθηκε με συντριπτική πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο. Νομίζω λοιπόν, αν αυτό το δούμε ως ένα εγκεκριμένο κείμενο, αυτό είναι σωστό. Και το λέω αυτό γιατί μερικές φορές τίθεται το θέμα του ορισμού των ε, καταγγελόντων. Ε, υπάρχει το κείμενο αυτό που έχουμε θετήσει και δεν νομίζω ότι πρέπει να ξαναξεκινήσει από αυτού του θέματος η συζήτηση από την αρχή. Για τις τροπολογίες που κατέθεσα, αυτές ε, είναι κατά λέξη αντιγραφή του ψηφίσματος. Αυτά που είπα εγώ ε, είναι γενικές τοποθετήσεις που έχει ήδη δεχτεί το Κοινοβούλιο και το, νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό είναι και πολύ πιο εύκολο να καταλήξουμε σε συμβασμό σε αυτήν την Επιτροπή. Και κάτι καινούριο στην Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμών ο ίδιος ο Ευρωπαίος ε, διαμεσολαβητής ή διαμεσολαβήτρια προφανώς έχει καταστήσει σαφές ότι με μεγάλη της χαρά να συμβάλλει και αυτή σε αυτό που χαρακτηρίζουμε ως ένα συμβουλευτικό φορέα για τους καταγγέλλοντες. Ε, προτιμοποιήθηκε να το κοιτάξει και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ξέρω ότι πολλοί συνάδελφοι λένε «Α, τώρα άλλος ένας ευρωπαϊκός οργανισμός, ανεξάρτητος, πολυγραφειοκρατία». Αν δείτε όμως ε, το ότι εδώ η διαμεσολαβήτρια μπορεί να βοηθήσει, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και εγώ σε μία από τις ε, τροπολογίες μου ακριβώς επισημαίνω και το ρόλο της διαμεσολαβήτριας, του διαμεσολαβητή γενικά ως θεσμού σε αυτή την υπόθεση. Κατά τα άλλα παραμένω σε αυτά που έχουμε συμφωνήσει και χαίρομαι πολύ που η κυρία Μακοβέη αναφέρθηκε στην ε, ερευνητική δημοσιογραφία γιατί αν δείτε ε, το κείμενο της σχετικής οδηγίας ε, και για του ε, καταγγέλντες και για την ερευνητική δημοσιογραφία δεν υπάρχει πολύ περιθώριο προστασία στην οδηγία. Γι' αυτόν ακριβώ το λόγο χρειαζόμαστε μεγαλύτερη προστασία και για τους ε, καταγγέλντες και βεβαίως για την ερευνητική δημοσιογραφία. Η Μπάρμπαρα. Πρόεδρε, Η προστασία των καταγγελόντων είναι απολύτως απαραίτητη. Αλλά θα πρέπει να περιορίζεται και να εστιάζει στο να αποφεύγει επαγγελματικές εμπλοκές που μπορεί να προκύψουν στην επαγγελματική ζωή δηλαδή ε, του ανθρώπου ο οποίος καταγγέλει. Ο τίτλος κάνει λόγο για καταγγέλλοντες οι οποίοι εργάζονται προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος. Όμως εκεί είναι λίγο δύσκολο να καταλάβει κανείς πότε ένας καταγγέλων εργάζεται προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος και πότε όχι. Έχουμε πολλές, πολλές ψευδείς ειδήσει τελευταία. Και πολλές τέτοιες καταγγελίες δεν προέρχονται τόσο πολύ ε, από μια διάθεση να ωφελήσουν οι καταγγελίες των δημόσιο συμφέρον, αλλά ίσως από μια διάθεση εκδίκησης ε, σε, έναν, σε ένα πρώην αφεντικό ή σε ένα συγκεκριμένο όργανο θεσμό κλπ. Και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την περίπτωση καταγγελιών που είναι ψευδείς. Σε αυτή την περίπτωση οι καταγγελόντες θα πρέπει να υφίστανται τις κατάλληλες ε, κυρώσεις. Όταν για παράδειγμα συκοφαντούν ή αμαυρώνουν τη φήμη κάποιου. Δημόσιο συμφέρον. Το δημόσιο συμφέρον μπορεί να έχει σχέση με την τρομοκρατία, με την άμυνα, ε, με την καταπολέμηση του οργανωμένου κλίματος κλπ. Είναι τομείς πολύ ευαίσθητοι και θα πρέπει να είμαστε και πολύ προσεκτικοί. Συνάδελφος από το σοσιαλιστικό, σοσιαλιστική ομάδα ανέφερε πως θα πρέπει ε, να δημιουργηθεί ένα γραφείο που θα βοηθάει ε, τους ε, καταγγέλλοντες με ή ε, θηγατρικές ή υποκαταστήματα ή τεσπρανογραφία σε όλη την Ευρώπη. Ήδη έχουμε πολλά προβλήματα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Μην προσθέσουμε και κάτι τέτοιο. Ίσως αυτό θα μπορούσε να ενταχθεί στα καθήκοντα του Ευρωπαίου Εισαγγελέα. Ευχαριστώ. Κατερίνα Τσινίτσι τώρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ πιστεύω μάλλον να το πω αλλιώς, προσπάθησα και εγώ να συμβάλλω με τις ε, τροπολογίες μου και τώρα θεωρώ ότι είναι απαραίτητο σε ευρωπαϊκό επίπεδο να έχουμε ένα νομοθετικό κείμενο το οποίο ε, θα ορίζει ε, το ρόλο των καταγγελόντων κυρίως στην αποκάλυψη διασυνοριακών φορολογικών υποθέσεων. Αυτά όλα είναι εγκλήματα, αυτά και άλλα που όπως σας είπα έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα. Χαίρομαι που ο συνάδελφος παρέθεσε ένα ψήφισμα ε, το οποίο θα μπορούσε να είναι και για μας ένα σημείο αναφοράς για να μπορέσουμε να ε, εργαστούμε, να προβάλλουμε, να στηρίξουμε το ρόλο των καταγγελόντων. Κατά την άποψή μου ε, δεν θα πρέπει να υπάρχει προστασία μόνο μέσα από νομοθετικές διατάξεις, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και μια ουσιαστική πολιτιστική αλλαγή. Να αναγνωριστεί ο ρόλος αυτών των πολιτών, γιατί αυτοί ε, πολλές φορές δεν περιορίζονται μόνο στα φορολογικά αλλά και σε άλλα θέματα επεκτείνονται ε, για τα θεμελιώδη δικαιώματα, για το περιβάλλον, για οτιδήποτε. Ε, βεβαίως και εγώ προσπάθησα να συνεισφέρω, όπως σας είπα, με τις ε, τροπολογίες μου θεωρώ ότι είναι σημαντικό οι αρμόδιες αρχές να μην αποκαλύπτουν την ταυτότητα των καταγγελόντων, ούτε και τις πληροφορίες που αποκόμισαν από αυτούς, γιατί μπορεί να προκύψει εκβιασμός εις βάρος τους. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το αναλύσουμε περαιτέρω, δηλαδή να υπάρχουν νόμιμες δίωδοι μέσα από τις οποίες οι καταγγέλντες... θα μπορούσαν να επισημαίνουν περιπτώσεις παρατυπιών. Η έκθεση αυτή με τις ε, απαραίτητες αλλαγές θα μπορούσε να οδηγήσει ε, σε σημαντικές ε, έρευνες και κατά την άποψή μου αυτό που παίζει ρόλο είναι στους καταγγέλλοντες να διασφαλίσουμε εγγυήσεις για τα δικαιώματά τους. Και βεβαίως και αν έχουν ζημιωθεί, αν ζημιωθούν από εκθεσμούς, να μπορούν να αποζημιώνονται. Σίγουρα σε αυτό το κείμενο πρέπει ακόμα να δουλέψουμε. Εγώ είμαι πρόθυμη να συμβάλλω, αλλά πιστεύω ότι είναι ένα σημαντικό κείμενο και θα πρέπει να ασχοληθούμε με το κείμενο αυτό, να το ορίσουμε και να το διευκρινίσουμε ακόμα περισσότερο. Ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Μέλλο, δεν είμαι σίγουρος ότι η κυρία Μακοβέη με κατάλαβε καλά αν κάποιος εργάζεται σε ένα όργανο και θέλει να καταγγείλει κάποια γεγονότα. παράδειγμα, δόθηκε μια εντολή και είναι τμήμα αυτής της πράξης και είναι τμήμα, λέω, έχει συμμετάσχει, έχει εμπλοκεί σε αυτή την πράξη πρέπει να προστατεύεται ή όχι. Δεν μιλώ για κάποιον ο οποίος έχει ήδη καταδικαστεί, μιλώ για κάποιον ο οποίος, έχει, οποίος εργάζεται σε ένα όργανο, σε μια εταιρεία κλπ. Παίρνει μια εντολή, θεωρεί ότι δεν είναι ορθή και φοβάται ότι αν καταγγείλει την εντολή αυτή μπορεί να θεωρηθεί και αυτός ο συνεργός. Τι θα γίνει με αυτόν. Πρέπει να προστατευτεί ή όχι. Δεν είναι καταδικασμένος ακόμα. Και αν εσείς είστε ο εισαγγελέας, ίσως εγώ θα ήθελα να πω έκανα το χ ψ δεν είμαι σίγουρος αν έδρασε σωστά ή όχι, θέλω όμως να το καταγγείλω αν με προστατεύσεις. Αν αυτούς δεν τους προστατεύσουμε, τους αφήσουμε εκτός του πεδίου εφαρμογή, τότε πολλά από πολλές τέτοιες πράξεις δεν θα διαρευνηθούν, διότι δεν θα καταγγελθούν οι άνθρωποι θα φοβηθούν. Δεν μιλούσα για καταδικασμένους. Δεν μιλούσα για κατάδικους. Μιλούσα για το πού ξεκινάει και πού τελειώνει η προστασία των καταγγελόντων. Εντάξει. Ε, η, η συγκήτρια για ορισμένα συμπεράσματα ενδεχομένω. Ναι, σας άκουσα με πάρα πολύ προσοχή. αλλάζει η εποχή και αυτή η συζήτηση το επιβεβαιώνει. Γιατί από τον κώδικα του Αμπουράμπη ε, μέχρι εδώ έχουμε, ε, ε, συζητούμε πάντοτε τα ίδια θέματα με διαφορετικό τρόπο. Το ψεύδος, πώς ξεχωρίζουν το ψεύδος από την αλήθεια. μόνο που τώρα έχει αλλάξει τεχνολογία, έχουν αλλάξει καιροί και όπως είπατε κι εσείς ε, η ψευδής καταγγελία, η ψευδορκία δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί ούτε να προστατευθεί. Και προφανώς ένα από τα στοιχεία τα οποία θα μας βοηθήσει στην αναζήτηση συνενέσεων είναι, η... είναι το τι εμείς μπορούμε ε, με βάση την δική μας εμπειρία και ε, εξειδίκευση να προσφέρουμε στην ε, Επιτροπή που είναι αρμόδια ε, επί της ουσίας. Υπάρχουν ορισμένα δικήματα και κάποια διασυνοριακά χαρακτηριστικά τους που μας υποχρεώνουν να αναζητήσουμε την αναλογικότητα αλλά και την αυστηρότητα της εργασίες μας, της σχολαστικότητα της εργασίες μας. Σημείωσα όλα όσα μας είπατε. Ε, όλα όσα αναφέρατε για, την για τη δική σας πρακτική εμπειρία, τους ε, ποινικού κώδικες που γνωρίζετε κλπ. Και από αύριο θα ξεκινήσω να δουλεύω τις ε, συμβαστικές προτάσεις. Για να βάλουμε και εμείς το δικό μας λιθαράκι ε, στο κείμενο της Επιτροπής Γιούρη. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα σας τα σχόλια. Thank you very much, Maita, and for everyone who took part in that debate. It was very good. Thank you. Um... Ευχαριστώ πολύ. Περιμένουμε μέχρι τις 5 η ώρα να, για να ξεκινήσουμε με την σεξουαλική κατεκοπή των παιδιών. Η εισηγήτρια δεν είναι εδώ ακόμα, ας περιμένουμε 10 λεπτάκια. Μια μικρή διακοπή λοιπόν μέχρι τις 5, παρακαλώ. Αλλά 5 ώρα ακριβώς παρακαλώ, ε. So 5 o'clock for point 18. Thank you. Um, Συνάδελφοι, θα ξεκινήσουμε. Η Άννα Μαρία έχει φτάσει. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν γιατί έχουμε και ψηφοφορίες μετά. Θέλω να γίνει ουσιαστική συζήτηση για σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ τους συναδέλφους που έχουν έρθει ήδη από τώρα. Υπενθυμίζω ότι είχαμε ψήφισμα στις 11 Μαρτίου για την ε, επιγραμμική σεξουαλική κακοποίηση και το Κοινοβούλιο ανέθεσε στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ να παρακολουθήσει περαιτέρω την ε, σχετική ε, οδηγία 2011-93 της Ευρωπαϊκής Ένωσης της οποίας η προθεσμία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο έληξε πρόσφατα. Πρόκειται λοιπόν για την έκθεση σχετικά με την ε, καταπολέμηση σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής τη παιδιών και τη παιδική πορνογραφία. Εμεί ζητήσαμε μία ε, μελέτη. Στις 25 Απριλίου κάναμε και ε, δημοσία για αυτό το θέμα. Υπήρξε και εσωτερική αξιολόγηση αντικτύπου για την υλοποίηση της οδηγίας. Θα ακούσουμε τώρα την παρουσίαση της έκθεσης τη ε, της συγκεκριάς μας Κοράτσα Μπίλτ Μπορούμε να δώσουμε το λόγο στην Άννα Μαρία να κάνει την παρουσίασή τη. Σε ευχαριστώ πολύ, Κλοντ. Σα ευχαριστώ όλου που είστε εδώ. Θα θυμάστε ότι και στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία ασχοληθήκαμε με αυτή την ε, ιστορική έκθεση, γιατί πράγματι επιτύχαμε ε, ελάχιστα ξεκάθαρα πρότυπα, ορισμούς και κυρώσεις, μέτρα για την ε, αποφυγή και καταπολέμηση του φαινομένου και προστασία των θυμάτων. υπάρχει λόγος ικανοποίησης αλλά και ε, υπάρχουν και ανησυχίες. Πρέπει να ασκήσουμε πίεση στα κράτη-μέλη για να συνεχίσουν ε, την ε, υλοποίηση και εφαρμογή της Οδηγία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή για τι δύο εκθέσει που, που έκαναν ιδίω για τη μεταφορά τη οδηγία στο εθνικό δίκαιο. Αναγνωρίζω και τι τεχνικέ δυσκολίε που αντιμετώπισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, για να συγκεντρώσει πληροφορίε από τα κράτη-μέλη. Όπως και να έχει όμω ε, πρέπει να μα πει μερικά πράγματα παραπάνω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πώ έχουν ε, εφαρμόσει την ομοθεσία τα κράτη-μέλη. Έχουμε βασιστεί σε μία ιδιαίτερα λεπτομερή ανάλυση ε, της ε, ερευνητικής υπηρεσίας, της υπηρεσίας ερευνών μάλλον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του EPRS και τους ευχαριστώ. Ε, είχαμε και τρεις δημόσιες ακροάσεις, Europol, Interpol, εμπειρογνώμονες της κοινωνίας των πολιτών, γραμμές υποστήριξης, ενδιαφέροντα μέρη, εισαγγελείς, από τα κράτη-μέλη, από όλο το φάσμα όσων ε, από την ε, πρώτη γραμμή ασχολούνται ε, με την καταπολέμηση αυτού του φαινομένου και με την προστασία των ανηλίκων. Αντίστοιχα είχαμε και συναδέλφους από τις ΗΠΑ και χαίρομαι που κάναμε τόσο καλή δουλειά, τουλάχιστον στο Κοινοβούλιο, για την προετοιμασία της εκθεσής μας. Έχουμε προσδιορίσει κάποιες ε, σημαντικές αδυναμίες ό,τι αφορά την εφαρμογή της οδηγίας και προτείνουμε συγκεκριμένες συστάσεις προς τα κράτη-μέλη ε, για την βελτίωση της ε, εφαρμογής. Τα σφάλματα, συγγνώμη, οι τομείς παρέμβασης είναι η δίωξη, πρόληψη, αρρωγή προς τα θύματα και η άρση ε, των εμποδίων για το περίφημο άρθρο 55. Θα περάσω στις ε, παρατηρήσεις, γιατί προσπαθήσαμε να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι. Σε ό,τι αφορά το ποινικό δίκαιο, καλούμε τα κράτη-μέλη να ενισχύσουν τις διατάξεις για την ε, σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων με όλες τις μορφές να εξετάσουμε μέτρα για τα δικήματα που αφορούν την σεξουαλική κακοποίηση από ενήλικες που έχουν ε, ε, πρόσβαση, που βρίσκονται σε κοντά δηλαδή σε ανηλίκους. Πρόκειται για δικήματα τα οποία διαπράττονται και στο διαδίκτυο ε, και εκτός. Πολύ συχνά όμως διαπράττονται από ενήλικες που γνωρίζουν τους ανηλίκους ή έχουν ε, θέση εξουσίας. Πρέπει λοιπόν ε, να διασφαλίσουμε ε, τη λογοδοσία, γιατί πολύ συχνά υπάρχει έλλειψη εποπτείας. Αναγνωρίζουμε ότι από το 2011 μέχρι τώρα υπάρχουν και νέες μορφές εγκλήματος, ιδίως στο διαδίκτυο, όπου πλήττει μια ολόκληρη γενιά, ιδίως τα κορίτσια σε αυτή την περίπτωση, με σεξουαλικό εκβιασμό και ε, συγκεκριμένες μορφές ε, σεξουαλικής παρενόχλησης, όπως είναι η χρήση της πορνογραφίας ε, ως εκδίκηση και έχει οδηγήσει και σε πολλές αυτοκτονίες. Καλούμε επίσης τα κράτη-μέλη να επεκτείνουν την, προθεσμία για την παραγραφή αυτών των δικημάτων για να, τα, για να διώκονται πραγματικά. Κάποιες φορές μπορεί να γίνει δίωξη πολλά χρόνια μετά την διάπραξη του δικήματο. Οπότε θέλουμε να ξεκινήσει αυτή η προθεσμία τουλάχιστον από τη στιγμή που τα θύματα ε, ενηλικιώνονται και μετά. Να ενισχυθεί η συνεργασία και να αξιοποιήσουμε υφιστάμενα εργαλεία όπως είναι το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Ερευνών και σύλληψη. Η Europol, η Eurojust θα πρέπει να ενισχυθούν ε, για να καταπολεμήσουν εγκληματικά δίκτυα, γιατί συχνά ε, πρόκειται για διασυνοριακές διαδικασίε. Πρέπει να δώσουμε στη Europol και στη Eurojust του κατάλληλους πόρους και εδώ θα, θα ήθελα ε, να ε, τις συγχαρώ αυτές τις δύο υπηρεσίες για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν και να υπάρχει και ανταλλαγή των πρακτικών σε ό,τι αφορά τι ερευνητικέ μεθόδου. Η ιδιαίτερη μνήμη πρέπει να γίνει ε, στην κατάσταση των ασυνόδευτων ανηλίκων και των ανηλίκων μεταναστών. Είναι μία από τις ε, απαράδεκτες εξελίξει που έχουμε δει μετά την ε, υιοθέτηση της οδηγία, γιατί είναι ιδιαίτερα ευάλωτα αυτά τα παιδιά στην διακίνηση, την σεξουαλική εκμετάλλευση και πρέπει να ενισχύσουμε την συνεργασία των αστυνομικών αρχών, τη διαλειτουργικότητα ε, των ε, βάσεων δεδομένων και το καθεξής. Μετά, πρόληψη. Ζητούμε από τα κράτη-μέλη ε, να θεσπίσουν μέτρα πρόληψης και παρέμβασης για όλα τα διαφερόμενα μέρη που έρχονται σε επαφή με παιδιά. Έχουμε συμπεριλάβει στο πακέτο για το άσυλο, για παράδειγμα, κατάρτιση για τους κυδεμόνες ε, των ασυνόδευτων ανηλίκων ή και η υποχρεωτική, υποχρεωτικός έλεγχος για τα άτομα που έρχονται σε επαφή με ανηλίκους, από καθηγητές μέχρι ε, Και πάλι να έχουμε ε, συλλογή ε, δεδομένων σε εθνικές βάσεις. Μετά, συνδρομή και προστασία των θυμάτων. Εδώ πρώτα απ' όλα θα ήθελα ε, να κάνω ιδιαίτερη μνήμα στην καταπληκτική δουλειά που γίνεται στην κοινωνία των πολιτών. Όλοι μας λένε ότι η συνεργασία με την κοινότητα των πολιτών είναι κρίσιμη σημασίας και Ξέρουμε ότι ε, τα παιδιά δεν εμπιστεύονται τόσο εύκολα έναν αστυνομικό, ενώ ε, οι μη όχι οι των πολιτών έχουν μια μεγαλύτερη ευκολία να προσεγγίσουν τα παιδιά, να εντοπίσουν τα θύματα, να κερδίσουν την εμπιστοσύνη τους και μετά ε, να μεταφέρουν την υπόθεση στις αρχές επιβολής του νόμου. Όμως κάνουν πολύ καλή δουλειά σε ό,τι αφορά τον εντοπισμό του επιγραμμικού υλικού. Για τη συνδρομή λοιπόν των θυμάτων καλούμε τα κράτη-μέλη ε, να ανταλλάσσουν τι πρακτικές για τα μέτρα προστασίας των θυμάτων, να αποφεύγεται η διπλή ε, θυματοποίηση και εδώ θα ήθελα να αναφερθώ ε, σε μια περίπτωση στη Σουηδία. Είχαμε και προσκεκλημένους από τη Σουηδία που είχαν ένα ειδικό πρόγραμμα προστασίας θυμάτων, ένα πολύ καλό παράδειγμα. Και βέβαια έχουμε και την σχετική οδηγία. τέλο κατάργηση ή κεφραγή τη πρόσβαση, Το άρθρο 25. Μόλι τα μισά κράτη-μέλη έχουν μεταφέρει το άρθρο 25 στην Εθνική Νομοθεσία. Αυτό είναι πολύ λυπηρό γιατί αυτό θα μας ε, επέτρεπε να ε, ε, φράξουμε την πρόσβαση ε, σε τέτοιες ε, φωτογραφίες στο διαδίκτυο. Πρέπει λοιπόν να εφαρμοστεί το άρθρο 25 και να μπλοκάρετε το περιεχόμενο στο διαδίκτυο το οποίο περιλαμβάνει παιδική πορνογραφία. Υπάρχει κατεπίγουσα ανάγκη να επιταχύνουμε τις διαδικασίες ε, απόσυρσης αυτού του υλικού από το διαδίκτυο ανεξάρτητα και από την αρχή της ε, αναλογικότητας. Και θα θέλαμε να εξετάσουμε και τη δυνατότητα του quick freeze, της ταχύτατας δηλαδή φραγής, ε, για να υπάρχει ένας επικαιροποιημένος κατάλογος ιστοσελίδων, γιατί υπάρχουν κάποιες ε, αποτρόπες ιστοσελίδες που εξακολουθούν να υπάρχουν, θα έπρεπε μέσα σε μερικές ώρες να κατεβαίνουν αυτές οι σελίδες. Και μετά τα κάτι μέλη ε, να μοιράζονται τους καταλόγους της μαύρης λίστας τέτοιων ιστοτόπων, και με την Interpol. Πρέπει να ενισχυθεί λοιπόν και ε, ο διαρθρωτικός διάλογος που κάνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είναι πολύ σημαντικός και η επένδυση στην τεχνολογία από τον κλάδο για την πλατφόρμα. Και εδώ, συναδελφέ, έχω αναφέρει ότι η τεχνολογία αναπτύσσεται και εξελίσσεται. Σαφώς και θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί σε αυτές τις τεχνολογικές εξελίξεις όλες αυτές οι τεχνολογίες θα πρέπει να ε, μας υποστηρίξουν. Ποτέ δεν πρόκειται να υποκαταστήσουν τον ρόλο της αστυνομίας και των αρχών επιβολής του νόμου. Πρέπει όμως να αξιοποιήσουμε όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Και να κάνουμε μία διάταξη, ούτως ώστε να είναι υποχρεωτικό για τους παρόχους ε, υπηρεσιών στη διαδίκτυο να καταγγέλουν τις περιπτώσεις ε, παιδικής πονογραφία, να ενισχύσουμε τον ρόλο ε, των τηλεφωνικών γραμμών υποστήριξη και να δώσουμε του κατάλληλου πόρου. Θα μείνω εδώ, Πρόεδρε. Περιμένω να ακούσω κατά σχόλια των συναδέλφων. Θα ήθελα μόνο να πω ότι όλοι θα πρέπει να αναλάβουν μερίδια της ευθύνης. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε, Αναμαρία, για αυτή την εισαγωγή. 30 λεπτά είχαν προβλεφθεί για αυτό το θέμα και είναι δική μου ευθύνη. Ζητώ συγγνώμη, δεν φτάνουν. Έχουμε στις 5.30 ε, δύο μεγάλες ε, ψηφοφορίες. Ε, Βεβαίω έχουμε εδώ δύο σκιώδεις εισηγητέ από τους σοσιαλδημοκράτες και τους Φιλεύθερους... Θέλει κάποιος άλλος να μιλήσει. Η Κατερίνα, κάποιος άλλος παρακαλώ. Εντάξει, τότε τρεις θα μιλήσουν, οι δύο εισηγητές και η Κατερίνα. Ε, και κανείς άλλος παρακαλώ. Γιατί πραγματικά πρέπει να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία στις 5.30 και πριν από την ψηφοφορία θα πρέπει ε, να έχει μιλήσει και η συγκήτρια η Μαρία. Ευχαριστώ ε, πρόεδρε, ε, χαιρετίζω την έκθεση της κυρίας Κορατσαμπίλτ. Ε, συμφωνώ με αυτά τα θέματα που αναφέρονται και επίση και αυτά που αναφέρει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αντιμετωπιστεί η σεξουαλική κακοποίηση κυρίως στο διαδίκτυο. Να σας πω και τη δική μας θέση. Πρώτα απ' όλα θα θέλαμε να επισημάνουμε κάτι το οποίο κατά την άποψή μας είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένα πορνογραφικό υλικό που να μην ισούται με σεξουαλική εκμετάλλευση. Έτσι πρέπει να το λέμε. Το να μιλάμε για παιδική πορνογραφία, αυτό είναι προσβολή. Στα χιλιάδες θύματα αυτού του ε, εγκλήματος, του αποτρόπαιου εγκλήματος οι γονικές οργανώσεις. Όλοι οι οργανώσεις θα πρέπει αυτό να το ονοματίζουν. Και μου έχουν ζητήσει τα θύματα της σεξουαλικής κακοποίησης που κάποια στιγμή η κακοποίηση αυτή μάλιστα επενέτηκε στο δικαστήριο μου ζήτησαν να τους δώσω μια φωνή, να τους υπερασπιστώ και να διασφαλίσουμε ότι η κακοποίηση τους αναφέρεται ως κακοποίηση και ως τίποτα άλλο. Αυτό ήταν το πρώτο. Το δεύτερο. Χαιρετίζω την έκθεση, αλλά αισθάνομαι ότι η έκθεση πρέπει γενικότερα να εξετάσει σημαντικά θέματα. Παραδείγματο χάρη, διαρωτώ με ε, ποιοι είναι οι συνοδοί των παιδιών που δεν έχουν άμεση σχέση με τα παιδιά, ε, παραδείγματος χάρη αυτοί που επεξεργάζονται προγράμματα ή ταξιδιωτικοί πράκτορες. Εγώ πιστεύω ότι όλοι όσοι έχουν σχέση με τα παιδιά, όλοι αυτοί θα πρέπει να αναζητείτε το ποινικό τους μητρό. Όλοι ανησυχούμε ε, σχετικά με τον ε, σεξουαλικό τουρισμό με παιδιά, αλλά ας είμαστε ξεκάθαροι. Αυτά γίνονται χωρίς να είναι ρυθμισμένα, γίνονται στην μαύρη κρυφή αγορά. Έτσι λοιπόν, κατά την άποψή μου, τον ε, αντιμετωπίζει αυτό το θέμα μόνο σε σχέση με τους αξιωτικούς πράκτορες, αυτό είναι το πρόβλημα. Το τρίτο, το να λέμε ένα κράτος μέλος πρέπει να βάζει φραγή σε ένα τέτοιο υλικό, αυτό δεν ικανοποιεί. Το υλικό παραμένει στο διαδίκτυο και ε, αυτό συμβάλλει στην κακοποίηση. Αν δεν ε, αφαιρείται γενικότερα το υλικό και αν αυτό δεν ε, τιμωρείται από το νόμο, τότε θα εξακολουθήσει η τιματοποίηση. Θα υπάρχουν τιμάτα, γιατί θα υπάρχει το υλικό και θα μπορούν οι άνθρωποι να το βλέπουν. Ως εκ τούτου δεν πρέπει να ε, αφαιρείται η φραγή. Αν θέλουμε να βοηθάμε τα θύματα, θα πρέπει να τους δίνουμε τη δυνατότητα να καταφύγουν στο κράτος δικαίου, που σημαίνει την ε, δίκη, διαδικασία δίκης και αποζημίωση. Ε, τα θύματα κατά την άποψή μας ε, τους αξίζει αυτό, τους αξίζει κάτι καλύτερο. Και τέλος, ε, τα θύματα είναι περισσότερα από τους δράστες. Εγώ λοιπόν θα ήθελα να υπάρξει μεγαλύτερη προσπάθεια για να βοηθηθούν τα θύματα. Και αυτό να γίνει, μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους, δηλαδή είναι η εξασφάλιση της ιδιωτικής του σφαίρας. Πρέπει, μπορούμε να δούμε τη Γερμανία. Εκεί μειώθηκε η προσφυγή στη, στα hotline ε, όταν ε, ε, πέρασε ο νόμος για την διακράτηση των στοιχείων. Δεν μπορούμε να καταλήγουμε σε μια κατάσταση όπου ε, τα θύματα δεν μπορούν να καταφύγουν σε αυτές τις ε, τηλεφωνικές γραμμές για να μιλήσουν γιατί φοβούνται ότι δεν διαφυλάσσεται η ιδιωτική τους σφαίρα. Ε, θα καταθέσουμε τροπολογίες και σε άλλα θέματα, αλλά ήθελα πρώτα απ' όλα να αναφέρω αυτά. Ευχαριστώ πολύ την εισηγήτρια για την έκθεσή της και ελπίζω ότι κατά τη διάρκεια των συναντήσεων των σκιωδών εισηγητών θα καταλήξουμε σε αποτελεσματικές συμβαστικές προτάσεις που θα λαμβάνουν υπόψη τους το συμφέρον των θυμάτων. Ε, κατάλαβα θα καταθέσετε και άλλες τυπολογίες, μας είπατε μόνο τα βασικά. Που αυτό ήταν πολύ καλό για σήμερα, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Σκαιώδης ε, εκ μέρους των φιλελευθέρων, η Νάταλη παρακαλώ. Ευχαριστώ, Κλοντ. Ε, ευχαριστούμε πολύ την Άννα Μαρία για αυτή την πολύ πλήρη εργασία της και ε, που δεν απέκλεισε τους και Ε, Είμαστε όλοι πεπισμένοι και προσιλωμένοι στον αγώνα αυτό και υπ' αυτή την έννοια είναι πολύ γλαφύρη ε, η δουλειά που έγινε από την Αναμαρία οδηγία αυτή είναι του 2011. Θα έπρεπε να έχει μεταγραφεί μέχρι το 2013. Πολλά όμως κράτη-μέλη δεν την έχουν ακόμα μεταγράψει. Η Κομισιόν αναφέρει ότι είναι περίπλοκη νομικά κλπ. Ωραία, εντάξει, αλλά εμείς δεν θεωρούμε φυσιολογική αυτή την καθυστέρηση και σίγουρα δεν μπορούμε να τη θεωρήσουμε αποδεκτή. Μιλούμε για ε, σεξουαλική κακοποίηση παιδιών. Και θα μπορούσαμε να είμαστε ακόμα πιο επικριτικοί, να μην περιοριστούμε μόνο στις, ε, ε, στην καταγραφή της κατάστασης. Νομίζω ότι μερικές φορές είμαστε πολύ διπλωματικοί και υπερβολικά ευγενικοί με την Κομισιόν. Καμιά φορά η Κομισιόν καθυστέρει μέχρι και ένα χρόνο να δημοσιεύσει εκθέσεις Στην ε, συνάντηση των σκιωδών συγκητών πολλοί είχαμε υπογραμμίσει πως δεν έχουμε καν αριθμητικά στοιχεία πάνω στο οποίο να βασίσουμε πραγματικά τις πολιτικές μας. Πιο συγκεκριμένα και εντάχει για τις τροπολογίες. Καταρχήν να πω ότι με ικανοποιούν όλες τις προσθήκες που έγιναν για πρόσθετα δικήματα. Επίσης χαίρομαι για τα όσα αναφέρονται για την πρόληψη άρθρα 21-24. Μία μόνο παρατήρηση ενδεχομένω. Ε, θα πρέπει ενδεχομένως να κάνουμε μία, ε, να, να από τα ορισμένες από τις προσθήκες που έγιναν γιατί αντιστοιχούν σε άλλη προβληματική. Ε, τώρα για το ε, για το γρήγορο πάγωμα ε, πιστεύω θα πρέπει να επιμείνουμε στη διαγραφή όχι στο πάγωμα. Και πρώτα θα πρέπει να μιλήσουμε τα κράτη-μέλη για τη διαγραφή και μετά για το πάγωμα. Αυτά σε γενικέ γραμμέ. Η έκθεση είναι πολύ καλή. Πιστεύω θα προχωρήσουμε γρήγορα. Thank you very much, Natalie. Katerina, could, uh, you, can ask just three Κατένα τρία λεπτά να έχει την καλοσύνη, γιατί πραγματικά μετά πρέπει να ψηφίσουμε. Πεντέμιση ακριβώ πρέπει να αρχίσει η ψηφοφορία. Ευχαριστώ, Κλώτ. Είναι πραγματικά πάρα πολύ σύντομη. Καταρχήν ευχαριστώ την συνάδελφο Κοράτσα Μπίλτ για τη δουλειά που έκανε για αυτή την έκθεση και εγώ ε, συμφωνώ μαζί σας όσον αφορά τα δικαιώματα των ε, ανηλίκων. Την ευχαριστώ λοιπόν για τη δουλειά τη ε, και εκείνη έχει προβάλει κάποια θέματα που είναι πολύ σημαντικά, Κυρίω το συντονισμό στο να συγκρίνονται αυτά τα εγκλήματα Συνέργεια λοιπόν, ε, Europol, Eurojust πρέπει να συνεργαστούν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και πρέπει ε, η συνεργασία να βελτιωθεί σε όλα τα επίπεδα. Κάτι άλλο που θεωρώ πολύ σημαντικό είναι να ε, προβλεφτούν νέες μορφές σεξουαλικής εκμετάλλευσης στο διαδίκτυο. Αυτά πλήττουν ε, κυρίως ε, τους ανήλικους και ευπρόσδεκτη είναι και η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών η οποία κοινωνία πρέπει να στηρίζει τους θεσμούς ε, για να αντιμετωπίζεται η σεξουαλική ε, κακοποίηση των ανηλίκων. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι το θέμα της ε, πρόληψης. Πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε σε αυτό το θέμα, σε όλα τα επίπεδα, να προβάλλουν τα δικαιώματα των ανηλίκων στο σχολείο, στην οικογένεια, στην κοινωνία των πολιτών, γιατί ξέρουμε ότι επειδή τα παιδιά καταφεύγουν περισσότερο στο διαδίκτυο, αντιμετωπίζουν όλους αυτούς τους ε, κινδύνους. Πρέπει και εγώ να πω ότι κατά την άποψή μου πρέπει να ε, δουλέψουμε πάνω σε ορισμένα θέματα. Αυτό το υπενήχθηκαν οι προλαλήσασες. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να δουλέψουμε ακόμα πάνω σε αυτό, γιατί ε, πρέπει να προβάλλεται λιγάκι το εμπόριο και η διάδοση πορνογραφικού υλικού με ανήλικα παιδιά. Κατά τα άλλα, όσον αφορά τη φραγή, και εγώ πιστεύω ότι πρέπει να δουλέψουμε πάνω σε αυτό, έτσι ώστε να καθίσετε δυνατό η επιγραμμική αφαίρεση του υλικού. Η προστασία των ανηλίκων. Κάτω από αυτό πρέπει, σας είπα, να εργαστούμε περισσότερο έτσι ώστε η ε, προστασία να είναι 100% η προστασία να αφορά τους ε, ανήλικους ε, οι οποίοι είναι θύματα της σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Αυτό που έχει επίσης σημασία είναι και η σεξουαλική εκμετάλλευση την οποία επίστανται τα ασυνόδευτα παιδιά μεταναστών. Ευχαριστούμε πολύ. Μαρία, δύο λεπτά σε παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν εξαιρετική η συνεργασία με όλους ε, τους σκιώδεις και θέλω να τους ευχαριστήσω, καθώς και τη γραμματεία και όλους ε, τους βοηθούς. Πολύ σύντομα, για την παιδική πορνογραφία, εγώ θα καταθέσω τροπολογία, γιατί δεν μπορούσαν να μπουν όλα αυτά τα στοιχεία στην έκθεση. Μεταξύ των πολλών τροπολογιών που θα καταθέσω θα έχω και μία για να αλλάξει η παιδική πονογραφία και να αποκαλείται πλέον σεξουαλική κακοποίηση. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε σε μία έκθεση πρωτοβουλία τον τίτλο τη οδηγία. Μπορούμε να κάνουμε όμω μια πολιτική μνήμα και θα δείτε ότι στη δική μου έκθεση πουθενά δεν υπάρχει διατύπωση παιδική πονογραφία». Μίριαν, επίση συμφωνώ μαζί σου, καθώς και με την Ναταλή και την Κατερίνα, ότι θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στην ε, ε, διαγραφή του υλικού και όχι στη φραγή του. Και θα προσπαθήσουμε να το ξεκαθαρίσουμε ακόμα περισσότερο στην ε, έκθεσή μου. Σα ευχαριστώ και για το Intergroup του οποίου προεδρεύω και εγώ και η Κατερίνα. Και εκεί πραγματικά υπάρχει το θέμα της μηδανικής ανοχής έναντι της ε, σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων ε, και της ατιμορρησίας. Αυτά τα δύο θέματα είναι θέματα προτεραιότητας για μας, και έχουμε κάνει σημαντική δουλειά και με την κοινότητα των πολιτών κατά τη διάρκεια αυτή τη θητείας Για την Επιτροπή, συμφωνώ ότι δεν είναι απαράδεκτη αυτή η καθυστέρηση. Γνωρίζουμε του λόγου. Προσπαθούμε στην έκθεση να είμαστε επικοδομητικοί, με το βλέμμα στραμμένο προς το μέλλον και ε, παρακαλούμε την Επιτροπή να ενημερώνει συστηματικά το Κοινοβούλιο και να μας ενημερώνει περισσότερο ε, σε σχέση με τη συμμόρφωση, με στατιστικά στοιχεία, ούτω ώστε το Κοινοβούλιο να συνεχίσει να ασχολείται με αυτό το ζήτημα με τον ε, στόχο της αυξανόμενης προστασία των ανηλίκων και πάντα στο πλαίσιο τη μηδενική ανοχή. Κλείνοντα, να πω ότι πρόκειται για πραγματικά ιδεχθή εγκλήματα τα οποία διαπράττονται σε βάρο των ανηλίκων, ακόμα ε, σε παιδιά ηλικία 2 ετών. Στην ε, έκθεση ε, υπήρχε ένας αστυνομικός στη Σουηδία για το ε, του τμήματος αγνοούμενων ανηλίκων που έλεγε ότι πρόκειται πραγματικά για παιδιά που είναι κάτω από 15 χρονών. Ένα ανήλικο έλεγε, κάποιο θα ήταν τόσο καλό μαζί μου, μου έδωσε που μου άφησε να κοιμηθώ στο σπίτι του, βέβαια έπρεπε να κοιμηθώ μαζί του. Και αυτό είναι ένα τρομερό τραύμα ε, που πραγματικά αφήνουν ε, ένα ανεξίτηλο σημάδι σε αυτά τα παιδιά. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μέχρι τις 18 Ιουλίου μπορείτε να καταθέσετε τροπολογίες. Ευχαριστώ πολύ. Θα ψηφίσουμε ακριβώς στις 5.30. Ε, και Καθίστε λοιπόν παρακαλώ και όλη η ψηφοφορία θα γίνει ηλεκτρονικά ως ήθιστε. Σε δύο λεπτά λοιπόν.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 Take your seats. They're too long votes, so... Παρακαλώ πολύ καθίστε. Έχουμε δύο ψηφοφορίες και πολυσέλιδες. Okay, everyone ready? Everyone isn't ready. Βάλε την κάρτα σου. Όλοι έτοιμοι. Ωραία. Όχι, ακόμα δεν είμαστε έτοιμοι. Παρακαλώ πολύ, καθίστε. Okay? Okay. Okay, colleagues, so the first... Πρώτη σοφορία. Πρώτο θέμα. Η συγγήτρια η κυρία Βόζενμπερκ. Κατά πολέμηση του κυβέρνου εγκλήματος. Αν δεν θέλει το λόγο η κυρία Βόζενμπερκ, μπορούμε να προχωρήσουμε στις ψηφοφορίες. Θέλετε το λόγο κυρία Βόζενμπερκ. Ε, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ Ήθελα να ευχαριστήσω τους σκιώδεις εισηγητές για την πολύ σημαντική δουλειά που κάναμε και τη συνεργασία που είχαμε, για την πληθώρα των ε, τροπολογιών που ήσαν συμβιβαστικές. Πιστεύω ότι θα δώσουμε μία, ένα μήνυμα, ένα πολιτικό μήνυμα μέσα από αυτή την έκθεση για το σκοπό που επιτελεί, για τον πόλεμο κατά του κυβερνοεγκλήματος. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Βόζεμπεργκ. Περνάμε στην ψηφοφορία. Έχουμε οκτώ προφορικέ τροπολογίε. Ξεκινάμε με την πρώτη, πρώτη τροπολογία. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Δεύτερη προφορική τροπολογία. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Τρίτη προφορική τροπολογία. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία υπαριθμών 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται προφορική τροπολογία υπαριθμών 5, άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 6, άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 7, άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 8. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1. Έναξη ψηφοφορία. Λήξη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Έναξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Άρχεται. Λίγη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 14. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 9. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 10. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 15. Ε, Μέχρι εκεί έχουν αποσυρθεί. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 16. Έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. 17. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. 18. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Τροπολογία. 19. Έναρξη λήξη, εγκρίνεται. Τροπολογία 20, έναρξη. Λήξη, εγκρίνεται. Τροπολογία 21, έναρξη. Λήξη, εγκρίνεται. Τροπολογία 22, έναρξη. Λήξη, εγκρίνεται. Τροπολογία 24. Έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. 25. Έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 1. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 26. Έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. 29. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. 32. Έναρξη. Λήξη εγκρίνεται. 33 έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. 34 έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 2 για την παράγραφο β του αιτιολογικού. Λίγη ψηφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 42. Έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 3. Εάν έρχεται η ψηφοφορία. Λίγη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 49. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 50. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 4. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Ανθρωπολογία 53, 56. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. 57. Έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. 58. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 5. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 6. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 66. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 7. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 75. Έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. 77. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. 78. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 8. Έναρξη. Λήξη εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 9. Έναρξη. Λήψη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 89. Έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. 90. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. 92. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. 93. Έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. 94. Έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. 96. Έναξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 10. Έναξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 11. Έναξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 12. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 109. Έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 13. Έναρξη. Έτσι. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 14. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 119. Έναρξη. 119 λέω. Λήξη. Εγκρίνεται. 128. Έναρξη. Λήξη. Απορρίφθηκε. 129. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Τροπολία 130. Έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. Τροπολογίες 131 και 132 που είναι ταυτόσιμες. Έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. Τροπολογία 133. Έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. 134 έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. 135 έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. 137 έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. 138. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται 147. Έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. 100, ε, συγγνώμη, ε, συμβαστική πρόταση 15. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 152. Έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. 153. Υπέρ. Ε, συγγνώμη, έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται.

Λήξη. Εγκρίνεται. 158. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. 159. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. 160. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. 163. Έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. 164. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. 165. Έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. 166. Έναρξη. Απορρίφθηκε ολοκληρωτικά. 167. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. 168. Έναρξη. Λήξη. Απορρίφθηκε. 169. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 16. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 175 έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. 176. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 17. Έναρξη. Εδώ ε, το ΕΛΚΑ έχει ένα παραπάνω, παρακαλώ να το διορθωθεί. Βέβαια, θα έχετε πάει καλύτερα σε σχέση με άλλες φορές και σας εγχαίρω. Μπράβο, Ρομπέρτα. Δεν ξέρω, με τηλεπάθεια <laughs> λειτουργείτε. Τώρα κλείνει λίγη ψηφοφορία, εγκρίνεται, δεν έχει και μεγάλη σημασία, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, συνάδελφοι, επιστρέφουμε στα δικά μας 1.85. Άρχεται. 1.85. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Απορρίτεται. Σημαντική 18. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 19. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 20. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. εγκρίνεται. Τροπολογία 203. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 204. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 205. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 207. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 208. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 21 άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 22. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 219. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 23. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 221. Παρακαλώ ψηφίστε. Πέρας. Απορρίπτεται. 223. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Να τις ε, εξετάσουμε από κοινού μέχρι την 228. 224 έως 228. Ναι σε όλα λέτε γιατί κοντεύει το καλοκαίρι, σας βλέπω. Λοιπόν, από κοινού 224 έως και 228 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται για λίγο. Σεβαστική 24. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε, εγκρίνεται. Στην ομιτοπολογία 234. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. 235. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 237. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 25. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 26. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. σοσιαλιστές ε, έκαναν κάποιο λάθος, οπότε πρέπει να επαναλάβουμε την ψηφοφορία. Δεν ξέρω τι ισχύει σύμφωνα με τους κανόνες, αλλά είμαι επίοικης λόγω θέρους. Λοιπόν, συμβαστική 26. Να ξαναψηφίσουμε την 26. Δεν υπερψηφίζουμε, όχι. Α, μάλλον εγώ ψήφισα λάθος. Α, αυτό δεν συμβαίνει συχνά. Οι στηρητικοί και οι μεταρρυθμιστές είναι συν ένας. Ευχαριστώ, Ντάνιελ. Βλέπω... Σε βλέπω ανακοφωσισμένο. Πέρας ψηφοφορία. Απορρίπτω. Λοιπόν, δύο 45. Μπριγκίτ, μην αρχίζεις, παρακαλώ. Λοιπόν, 2.45, όπως σας έλεγα. Πέρας. Απορρίπτεται. 2.46. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 2.47, 48 έως και 52. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. 2.53. Άρχεται. Α, συγγνώμη συνάδελφοι, έκανα λάθος. Σεβαστική 27. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Τροπολογία 270. Έναρξη. Πέρας. Απορρίπεται. 271. Έναρξη. Αφήνω ανοιχτή την ψηφοφορία, γιατί αλλάζετε θέσεις. 2,71 ακόμα συνεχίζει την ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 272. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 273. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. 274. Έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. 2.75. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 2.76 έως και 2.79 ταυτόσιμες. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 28. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 29. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 30. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 294. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 295. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 2.96. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 2.97. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 2.99. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Σημαντική 31. Άρχεται. Πέρασε. Εγκρίνεται. 303. Μάλλον 304. Όχι, 303. Έναρξη. Πέρας. Οι σοσιαλιστές έχουν ένα παραπάνω εδώ. Μπριγκίτ, ένας παραπάνω από τους σοσιαλιστές. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 300. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 32, συνάδελφοι. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 33. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Σημαντική 34. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 322. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 303. Συγγνώμη, 323. Έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. 325-326 ταυτόσημες. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 329. Έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. 330. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 3.31. Έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. 332. Έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. 333. Έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. 334. Έναρξη. Θα μπορούσαμε να τις ψηφίσουμε από κοινού βέβαια. Πέρας. Απορρίπτεται. ταυτόσουμε σε 3.35-3.36. Έναρξη. Πέρας. Έγκρινατε. Συμβαστική 35. Έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. 3.38. Άρχεται. Πέρας. 3.38. Επαναλαμβάνει ο Πρόεδρος. Ψηφίσατε όλοι. Θα το ξανακάνουμε. Και αν βιάζομαι να μου το λέτε. Απλώ επειδή κανεί δεν μου λέει τίποτα, προχωράω. Ησυχία παρακαλώ, γιατί όταν ε, επικρατεί ησυχία πάμε πιο γρήγορα. 3.38, επαναλαμβάνουμε τη 3.38. Άρχεται. Ησυχία παρακαλώ, πέρας. Εγκρίνεται. 3.39. Ένα δεξί. Πέρας. Εγκρίνεται. 3.37. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 3.40. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 101. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 3.41. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 3.43, 3.44 ταυτόσιμες άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 3.45. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 3.46. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 3.47. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Από το ΕΛΚ υπάρχει ένας παραπάνω. Παρακαλώ να το διορθώσετε. Συμβαστική 36 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 37, Η 37, ψηφίζουμε παρακαλώ. συμβαστική 37, έκλεισε ψηφοφορία. Εγκρίνεται. ...3.70 και 3.71. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Η 372. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε. Απορρίπτεται. Τρία ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 358. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Όχι, δεν είναι 358, ρωτάει ο πρόεδρος. Συνάδελφοι, ε, ακυρώνεται αυτή η ψηφορία. Σα ευχαριστώ που ψηφίσατε, αλλά πάμε στην 349, για αυτήν έπρεπε να ψηφίσουμε. 349 και ζητώ συγγνώμη γιατί ήταν δικό μου το λάθο. Το 349, παρακαλώ, ψηφίζουμε. ...349, έκλειση ψηφοφορία, απορρίπτεται. Η συμβαστική 38, ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Η 373. Ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 374 και 375 ταυτόσιμες ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Για 376 ψηφίζουμε. Έκλειση ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 377 ψηφίζουμε. Έκλεισε. Εγκρίνεται. 378 Έκλεισε. Απορρίπτεται. 381, 382, ταυτόσιμες ψηφίζουμε. Έκλεισε. Απορρίπτεται. 383, ψηφίζουμε. Έκλεισε. Απορρίπτεται. 384. Ψηφίζουμε. Έκλεισε. Εγκρίνεται. 386 και 387 ταυτόσημες ψηφίζουμε. Έκλεισε. Απορρίπτεται. 388 ψηφίζουμε. Έκλεισε. Απορρίπτεται. 389. Έκλεισε. Απορρίπτεται. σημειβαστική 39. Έκλεισε. Εγκρίνεται. σημειβαστική 40. Ψηφίζουμε. Έκλεισε. Εγκρίνεται. 396 ψηφίζουμε. Έκλεισε. Εγκρίνεται. 397. Έκλεισε. Απορρίπτεται. 398. Ψηφίζουμε. Έκλεισε. Απορρίπτεται. 399. Έκλεισε. Απορρίπτεται. Η 400 Έκλεισε. Απορρίπτεται. Η 41. Εγκρίνεται. Η 406. Ψηφίζουμε. Έκλεισε. Απορρίπτεται. Η 405. Ψηφίζουμε. Έκλεισε. Εγκρίνεται. 401. Έκλεισε. Εγκρίνεται. 402. Ψηφίζουμε. Έκλεισε απορρίπτεται 404 έκλεισε εγκρίνεται 407 και 408 ταυτόσιμες ψηφίζουμε έκλεισε απορρίπτεται 409 Έκλεισε. Απορρίπτεται. Τελειώσαμε σχεδόν. 4-10. Ψηφίζουμε. Έκλεισε. Απορρίπτεται. 4-1-1. Ψηφίζουμε. Γκρίνεται. 4-12. Ψηφίζουμε. Έκλεισε. Απορρίπτεται. Η συμβαστική 42. Ψηφίζουμε. Έκλεισε. Εγκρίνεται. 4-20. Ψηφίζουμε. Έκλεισε. Εγκρίνεται. 421. Ψηφίζουμε. Έκλεισε. Απορρίπτεται. 422. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε. Απορρίπτεται. 4.23 ψηφίζουμε. Έκλεισε. Εγκρίνεται. 4.25 ψηφίζουμε. Έκλεισε. Απορρίπτεται. 426 ψηφίζουμε. Έκλεισε. Εγκρίνεται. 427 ψηφίζουμε. Έκλεισε. Εγκρίνεται. 428, 429 ταυτόσημες, ψηφίζουμε. Έκλεισε. Απορρίπτεται. Η 4.30 ψηφίζουμε. Έκλεισε. Απορρίπτεται και τώρα ψηφίζουμε για το σύνολο του κειμένου ως ε, τροποποιήθηκε ε, και ψηφίζουμε παρακαλώ. Has everyone η ψηφοφορία. Συγχαρητήρια κυρία Βόζεμπεργκ. Συγχαρητήρια στην εισηγήτριά μας. Ευχαριστούμε συνάδελφοι για την ε, υπομονή σας. Ξέρω, για την πρώτη σας ευχαριστώ. Έχουμε κι άλλη να επιδείξετε πειθαρχία παρακαλώ και ηρεμία γιατί έχουμε και άλλη μια μεγάλη ψηφοφορία. Όχι, να ξεκινήσουμε. Yeah, keep, keep the vibe going. So colleagues, we uh, move quick. Let's just move fast onto all of them, okay? Λοιπόν, πάμε τώρα στην ε, στον προτινόμενο κανονισμό για τις άδειες παραμονής, εισηγητής ο κύριος Χαλαχάχου του ECR. Θέλετε να πείτε κάτι? Όχι, δεν θέλει να πει τίποτα. Ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε για το κείμενο που συμφωνήθηκε, στι στις ε, διοργανικές διαπραγματεύσεις. Ψηφίζουμε παρακαλώ. σε όλους περισσεύει ένας και στην ΚΟΕ περισσεύει ένας. Όχι το ECR, το ECR ε, περισσεύει, στο ECR περισσεύει ένας. Παρακαλώ ένας από το ECR να αφαιρέσει την κάρτα του για να ολοκληρώσουμε την ψηφοφορία. Σας παρακαλώ δεν γίνεται. Πρέπει, ε, παρακαλώ, η ΣΥΑΡ να αφαιρέσετε μία κάρτα για να ολοκληρώσουμε την ψηφοφορία. Είχαμε δύο που περίσευαν. Ωραία. Λοιπόν, τέλειωσε η ψηφοφορία. 52 υπέρ, 2 κατά, καμία αποχή. Συγχαρητήρια στον εισηγητή, τον κύριο Χαλαχάχο. Χαλαχάχο.